ενημέρωσαν σχετικά. Προχωρούμε λοιπόν, εγκρίνοντας την ημερήσια διάταξη, εφόσον συμφωνούν και οι συντονιστές. Επίσης, θα ήθελα να σας ζητήσω να εγκρίνουμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις 20 και 21 Ιουλίου. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις επί των πρακτικών, θα τα υπογράψω ως εγκριθέντα. Εντάξει, ευχαριστώ. Σημείο 3. Εδώ είναι ο κύριος Κόλιτσεκ. Α, δεν δεν Το σημείο 3 είναι η εξέταση του προπολογισμού του 2010 σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες. Κύριε Κόλιτσεκ, έχετε το, το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να σας ευχηθώ σε όλους και καινούριου και ανακυκλωμένους ευρωβουλευτές. Καλή επιστροφή. Και καλή τύχη. Ελπίζω ότι σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες θα συμφωνήσουμε επί των βασικών αρχών. Εγώ θα συνεχίσω τη δουλειά που ανέλαβα μέχρι τώρα και είμαι σίγουρος ότι θα θυμάστε ότι μου ανατέθηκε η ευθύνη της ε, ε έκθεσης, είμαι ο εισηγητής, αλλά δεν έχω τα στοιχεία, δεν μου δώσαν τα στοιχεία από το ε, Συμβούλιο και κατά συνέπεια οι τροπολογίες που έχετε λάβει ε, προσπαθούν να προτείνουν και να υποδείξουν ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να επανέλθει στις ε, παλαιότερες, στα παλαιότερα νούμερα. Να εξηγήσω τι θέλω να πω exaktní Η οικονομία προφανώς δεν είναι ακριβής επιστήμη και κατά συνέπεια κάθε οικονομολόγος έχει τη δική του απάντηση για την κρίση, αλλά όλοι συμφωνούν ότι σε περιοχές κρίσεων πρέπει να επενδύουμε σε μεγάλα έργα υποδομών. Οι περισσότερε γραμμέ του προπολογισμού στον προπολογισμό τη επιτροπή μα στον τομέα των μεταφορών δηλαδή, ακριβώς προς τα εκεί αποβλέπουν. Υποδομές μεταφορών. Υπάρχουν και άλλα θέματα, το ΕΑΣΑ για παράδειγμα, άλλες υπηρεσίες. Ωστόσο, οι γραμμές για τις δομές αυτές είναι χαμηλότερες σε σχέση με τις ε, επενδύσεις τους διάφορους διαδρόμους. του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Και προφανώς εν ώψη της αύξησης της, ε, μάλλον για να πετύχουμε αύξηση της απασχόλησης πρέπει να πετύχουμε αύξηση της ανάπτυξης. Στην προηγούμενη ε, θητεία ε, κατακρίθηκαν οι χαμηλές πιστώσεις που είχαν δοθεί για τις, τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Οι περισσότερες τροπολογίες, το 90% των τροπολογιών στον, στις ε, μεταφορές αυτό το στόχο έχουν. Θέλουμε να υπάρξει ή να επανέλθει το αρχικό ποσό που υπήρχε σε κάθε θέση τον, ε, του προπολογισμού για τις μεταφορές και για τον τουρισμό. Σε ό,τι αφορά τις λοιπές προτάσεις, πιστεύω ότι θα ήταν καλή ιδέα να εναρμονίσουμε την διατύπωση που χρησιμοποιούμε, Φερρυπίν, ε, στη γραμμή 6400 για τον τουρισμό η διατύπωση εκεί θα πρέπει να είναι πανομοιότυπη με τη διατύπωση που έχουμε σε άλλα τμήματα του κειμένου. Δηλαδή να, ενομοιώ, να, να εξομοιώσουμε τις, ε, ε, την οδολογία. Θα έπρεπε λοιπόν να επανεξετάσουμε στο σημείο αυτό τι κάνουμε. Έχουμε τρεις γραμμές. που θέλουμε να ανεβάσουμε. Και το ερώτημα είναι ξεκινούμε από το χαμηλότερο ποσό ή από το ψηλότερο ποσό. Νομίζω ότι υπάρχει μια καλή πρόταση για το Μάρκο Πόλο. Η 6416 της κυρίας Βόρτμαν Κόλ που θέλει να αυξήσει σημαντικά τα ποσά αυτά. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους γιατί τα σχόλιά της, τα σχόλιά τους ε, όπως βελτίωσαν την αρχική μου πρόταση. Θέλω εξ να ε, υπογραμμίσω ότι θα χρησιμεύσουν πάρα πολύ όταν ξεκινήσουμε τις ε, αψιμαχίες με την Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών που θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου. Πολύ θα ήθελα να δω πώς θα είναι η ατμόσφαιρα και δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να πείσουμε την Επιτροπή Προϋπολογισμών ότι σε περίοδους κρίσεων θα πρέπει να επενδύουμε σε μεταφορές η συνάδελφος κυρία Τικάου για παράδειγμα προτείνει να προχωρήσουμε όπως είχαμε με τον ίδιο τρόπο που είχαμε και στην προηγούμενη θητεία. Να εξετάσουμε την ε, πλωτή οδό στον ε, Δούναβη, νομίζω προστέθηκε στο κείμενο, και να εξετάσουμε κατά πόσον το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης θα μπορούσε να πάει σε, ένα άλλο, σε μια άλλη κατηγορία, σε ένα άλλο τμήμα του προπολογισμού, όχι στο τουρισμό και μεταφορές, διότι θυμάμαι ότι όταν συζητούσαμε το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, ε, είχε μπει ο τουρισμός και μεταφορές σε ένα τμήμα, ενώ τον Γαλιλαίο είχε πάει σε χωριστό, ήταν ξέχωρο, είχε πάει σε χωριστό τμήμα. Άρα ε, αυτό είναι ένα ζήτημα που θα ήθελα να συζητήσουμε. Θεωρείτε ότι το κεφάλαιο για τις μεταφορές θα έπρεπε να περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα ή θα έπρεπε τα προγράμματα αυτά να έχουν χωριστές γραμμές. Όταν το συζητήσουμε και αποφασίσουμε, εγώ θα έρθω για θα πάω για να αιτιολογήσω την επιλογή μας. Αυτά εισαγωγικά. Θέλω να σας πω ότι, ήμουν, ε, ότι είμαι πολύ ευτυχής που είδα ότι η έκθεση αυτή ξεκινά με βάση παρόμοιες θέσεις και πολλές τοπολογίες που ακριβώς το ίδιο στόχο έχουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κόλιτσεκ. Ο κύριος Γκρός για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση αυτή, γιατί άλλωστε οι θερινές διακοπές δεν είναι ο ιδανικός ε, χρόνος, αν θέλετε, για να κάνουμε τέτοιες εργασίες, αλλά νομίζω ότι πολλές, ε, πολλά σημεία συμφωνίας έχουμε βρει στην Επιτροπή. Να αναφέρουμε κάποια στοιχεία τώρα. Υποστηρίζουμε τις προτάσεις και σε μεγάλο βαθμό στις πρώτες προτάσεις που δεν έχουν περιοριστεί δηλαδή. Νομίζω ότι υπάρχει συνοχή τώρα σε ό,τι αφορά τις εποχές κρίσης. Συμφωνώ απόλυτα ότι όντως χρειάζονται αύξηση των επενδύσεων σε τέτοιες περιοχές χωρίς ε, επιπρόσθετες επιβαρύνσεις για την επόμενη γενιά. Και αυτό λοιπόν ισχύει ιδιαίτερα για τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Πρέπει πραγματικά να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπροστά. Και επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω και να πω ότι λυπάμαι επειδή σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της κρίσης δεν έχει εξοπλιστεί με τα απαραίτητα μέσα οι μεταφορές. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι που θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Θα πρέπει να βρούμε με τα ήδη φυστάμενα κονδύλια και να προωθήσουμε προγράμματα. Και νομίζω ότι στις μεταφορές μπορούμε να θέσουμε νέα έμφαση, ακόμα και σε εποχή κρίσης. Κάτι τέτοιο πραγματικά θα απαραίτητο και γι' αυτό λοιπόν ότι θα πρέπει με αποφασιστικότητα να ζητήσουμε από την Επιτροπή Προπολογισμών να θέσει αυτή την έμφαση. Κάτι άλλο. Πολύ συχνά συζητιέται στις θερινές διακοπές το καλοκαίρι τα θέματα προϋπολογισμού. Αλλά απαραίτητο θα ήταν να έχουν πιο πολλές πληροφορίες και οι βουλευτές. Για παράδειγμα για τη μείωση κάποιων εξόδων. Ότι υπάρχουν για παράδειγμα κάποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τη μείωση των εξόδων. Νομίζω ότι καλό θα ήταν και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας δοθούν πιο πολλές ε, πληροφορίες για την αξιοποίηση κάποιων κονδυλίων για κάποια πιλωτικά προγράμματα, γιατί από αυτό θα μπορούσαμε να μάθουμε, για παράδειγμα, σε θέματα συγχρηματοδότησης. Νομίζω ότι για μας ως βουλευτές είναι σημαντικό να ξέρουμε όχι μόνο πόσα κονδύλια έχουμε, αλλά και γιατί αξιοποιούνται ή ενδεχομένως γιατί δεν αξιοποιούνται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ύστερα αναφέρθηκαν και άλλα ζητήματα. Το θέμα της ασφάλειας είναι σημαντικό. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε τα κονδύλια και θα πρέπει να συνεχιστούν κάποια πολιτικά προγράμματα. Θα πρέπει να μπορέσουν να συνεχιστούν προγράμματα έρευνας. Έρευνας που αποσκοπεί σε πληροφορίες που θα βελτιώσουν την ασφάλεια. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να συνεχιστεί. Σε ό,τι αφορά το Μαρκοπόλο θα κοιτάξουμε τις ε, τροπολογίες και θα συντονιστούμε με τη συνάδελφο Βόρτμαν Κόλ προκειμένου να συντονίσουμε τις παρατηρήσεις μας και μια άλλη παρατήρηση του συναδέλφου, ο οποίος έκανε κάποια σχόλια σε ό,τι αφορά τον τουρισμό με το ποδήλατο. Και εγώ, και εμένα μου αρέσει το ποδήλατο, αλλά δεν ξέρω αν πραγματικά έχει να κάνει με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Και να πω ότι αν είναι διχασμένο το αποτέλεσμα στην ψηφοφορία εκ μέρου του ΕΛΚ, δεν έχει να κάνει τίποτα αυτό με το κατά πόσο μα αρέσει το το ή όχι. <laughs> Πολύ ευγενικό εκ μέρου σα. Σα ευχαριστούμε κύριε Γκρό, λέει ο πρόεδρο. Εκ μέρου των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών, ο κ. Αλικαντράουε. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Έχω την αίσθηση ότι σε γενικέ γραμμέ συμφωνούμε γενικά. Και εμεί υποστηρίζουμε τις περισσότερες από τις τροπολογίες οι οποίες αποσκοπούν στη διατήρηση τουλάχιστον του επίπεδου της χρηματοδότησης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ομάδα μου συμφωνεί απόλυτα ότι όντως σε εποχές κρίσης δεν μπορούμε να παριορίσουμε τα προγράμματα εκείνα που πραγματικά μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάκαψη. Και πραγματικά οι επενδύσεις στις μεταφορές δεν ε, σημαίνουν μόνο στο να επενδύουμε σε κάτι το οποίο σήμερα θα αποφέρει θέσεις εργασίας. Όχι. Σημαίνει και επενδύσεις για δυνατότητα ανάπτυξης στο μέλλον, για πιο βιώσιμα συστήματα μεταφορών. Όλα αυτά μπορούν να αποφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης στο μέλλον. Και γι' αυτό λοιπόν θα υποστηρίξουμε τις σχετικές προτάσεις του εισηγητή. Να ευχαριστήσουμε και τον εισηγητή για τις προσπάθειες και τη δουλειά που έκανε στους καλοκαιρινούς μήνες. Κάποιες ε, τροπολογίες που είναι πιο φιλόδοξες θα πρέπει να τις, να τις εξετάσουμε πιο λεπτομερώς, αλλά νομίζω ότι πραγματικά σε γενικές γραμμές μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ. ο Στέρξ για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Είναι σαφές ότι και εμεί ακολουθούμε τη γραμμή του εισηγητή και τον ευχαριστούμε. Δεν είναι σήμερα η στιγμή να μειώσουμε τι προσπάθειε μα στον τομέα των μεταφορών. Θα πρέπει να διατηρήσουμε τουλάχιστον το επίπεδο που έχουμε πετύχει. Άρα θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο Γκρό. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στην Επιτροπή προπολογισμών ότι έχουμε ένα κατάτατο όριο, το οποίο δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε, δεν θέλουμε να πέσουμε κάτω το επίπεδο αυτό. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω. Αυτές οι λεπτομέρειες τις ακούσατε και από τους συναδέλφους. Thanks. Ευχαριστώ. Κυρία Λίχτεμπορή για τους πράσινους παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ με τη γενική αυτή γραμμή, αλλά αυτό που θα ήθελα σε κάθε περίπτωση να αναφέρω είναι τις προτεραιότητες που θα πρέπει να θέσουμε σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό. και μιλώ για τα δικαιώματα των ε, επιβατών και θεωρώ ότι είναι σημαντικές όλες οι σχετικές τροπολογίες που υποβλήθηκαν γιατί αυτό πραγματικά το περιμένει ο λαός της Ευρώπης από μας. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις διεθνείς μεταφορές. Να υπάρξει και οικονομική δέσμευση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεωρώ ότι αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί το σύστημα των δημοσίων μεταφορών αν θέλετε, είναι τόσο καλό όσο καλές είναι και οι υπηρεσίες που παρέχονται στους επιβάτες. Αν θέλουμε λοιπόν σε περίοδους κρίσης να επενδύσουμε στις μεταφορές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και την επερχόμενη συνάντηση στην Κοπεχάγη για το κλίμα, το θέμα λοιπόν είναι σε ποιους τομείς θα επενδύσουμε. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες. Πιστεύω λοιπόν ότι στο Μάρκο Πόλο και ότι το Μάρκο Πόλο και η έρευνα είναι η τομή εκείνη που είναι η που είναι πιο σημαντική. Για να μην προωθήσουμε δηλαδή μόνο τρόπους μεταφοράς οι οποίοι θα είναι επιβλαβείς προς το περιβάλλον. Και κάτι τελευταίο σε ό,τι αφορά του χρηματοδοτικούς πόρους για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και τη συγχρηματοδότηση. Είναι πολύ σημαντική από ψυχολογικής άποψης η συγχρηματοδότηση. Δεν είναι κάτι δηλαδή που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόκειται για ένα κοινά, από κοινού αναπτυγμένο πρόγραμμα. Γι' αυτό είναι λοιπόν τόσο σημαντική η συγχρηματοδότηση. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την χρηματοδότηση υποδομών σε κάποιες χώρες, δεν θα γίνει αποτεκτό αυτό και δεν θα προωθήσει και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε Υπάρχει αυτό το πρόβλημα με την ε, έλλειψη, αν θέλετε, συμμετοχής από τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι εμείς ως Επιτροπή θα πρέπει να πούμε ποιο είναι το πρόβλημα, ότι αφενός ε, οι αρχηγοί κυβερνήσεων αποφασίζουν να διαθέτουν όλο και λιγότερα κονδύλια σε προγράμματα συγχρηματοδότησης και μετά έρχονται και παραπονιούνται ότι δεν έχουν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ξεπερνάει, αν θέλετε, κάπως τις ε, τροπολογίες από πλευρός ε, προϋπολογισμού, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό γιατί δεν μπορούμε να αφήνουμε τα κάτι μελη να την βγάζουν, αν θέλετε, καθαρή με τέτοιε δικαιολογίε. Κύριε Ζήλα, παρακαλώ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα ε, ήθελα να πω κι εγώ, όπω είπε και ο προλαλή σα, και τι τροπολογίε τι οποίε είχε υποβάλει. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο και θα πω το εξή, ότι παρακολουθώ την, ακολουθούμε την ίδια γραμμή για αυτά τα οποία έλεξα μέχρι τούδε για αυτό το θέμα. Αλλά όσον αφορά τις δαπάνε και τις περικοπές που πρέπει να γίνουν θα πρέπει να προσμένουμε και θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Θα πρέπει να προσπαθώσουμε αυτή τη στιγμή να μην, να περάσουν πάρα πολλέ περικοπές κατά τομή. Αλλά βεβαίω, θα πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστέ και από την εμπειρία που έχω εγώ από τη χώρα μου Σήμερα εκεί ο, προπολογισμό έχει περικοπεί πάρα πολύ δραστικά. Αυτό είναι να δούμε πραγματικά ποια θα είναι και η μακροχρόνια και βραχυπρόθεσμη επίπτωση επί της οικονομίας επίσης. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να γύρω αυτή τη στιγμή βασικά είναι, δεν είναι πολύ εύκολη θέση, αλλά η συντηρητική πλευρά έχει την ίδια πρόταση την οποία έχουμε κάνει όπως και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λαμπρά. Αυτή τη στιγμή κλείνει κατά αυτόν τον τρόπο αυτή τη στιγμή ο κύκλο των συντονιστών. Δεν ξέρω πραγματικά αν κάποιο θέλει να πει κάτι, να προσθέσει. Α ε, επιδείξει το, Ο κύριο Μπράτπορν θέλει να πάρει το λόγο. Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έλεγα αυτή τη στιγμή πω κάτι όταν αυτόν τον κύριο Κόρτσεκ και αυτά τα οποία είπε προηγουμένω. Καθότι, τελική αναλύση, όταν δούμε τι τροπολογίε αυτή τη στιγμή την οποία έχουμε αναχείρα, εάν πραγματικά σκέπτεται και θέλει τελικά να βελτιώσει το δίκτυο των μεταφορών και θέλει κάτι αυτό το οποίο θα πρέπει να έχει όσον αφορά τις υποδομές και το πρόγραμμα το οποίο έχει υπάρχει όσον αφορά την προηγμό του ε, ε, θα πρέπει να δει την οικονομία σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Βεβαίω έχω μια συμπάθεια σε αυτό το θέμα. Πριν λοιπόν ακριβώς πρέπει κάνουμε οτιδήποτε, πρέπει να δούμε σπιθαμή προς σελίδα προς σελίδα, ποια είναι εκείνη η διοικητική διαχείριση η οποία γίνεται. Δεν είναι αυτή τη στιγμή τίποτα άλλο παρά μια διαχείριση διοικητική η οποία θα πρέπει να γίνει και δεν, δεν υπάρχει λοιπόν μια οποιαδήποτε επένδυση κεφαλαίων η οποία θα πρέπει να γίνει σε αυτό το πέρα. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο βλέπω προτάσεις οι οποίες έρχονται και οι οποίε θέλουν την αύξηση του κεφαλαίου αυτή τη στιγμή αυτής της εταιρεία η οποία ε, ασχολείται με αυτό το θέμα. Δεν είναι όμως πρόταση αυτή τη στιγμή η οποία υπάρχει μέσα σε αυτό το κείμενο το οποίο εξετάζουμε και το οποίο θα θέλαμε να υπάρχει μέσα στο προπολογισμό του ΕΕ. Εάν ακολουθήσουμε αυτό το, το μονοπάτι, αν θέλετε, αυτή το σκεπτικό, θα πρέπει να δούμε πραγματικά ποιο είναι η ασφάλεια η οποία παρέχεται και η ασφάλιση η οποία δίνεται και ορισμένες αξίες οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούν ώψιν ε. Αλλά όταν δω όλες τις τροπολογίες μία προς μία, σελίδα προς σελίδα, απλούστατα υπάρχει χρήματα τα οποία πάνε προς τη γραφειοκρατία παρά σε προγράμματα τα οποία είναι συγκεκριμένα και αυτά. Και εδώ πραγματικά σε τι χρησιμεύει αυτή η Επιτροπή. Γιατί αν παρακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι, αυτή την ατραπό, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν μέλη τα οποία και το έχουν πει και σε παλαιότερες εποχές ότι Υπάρχει ένα ολόκληρο στρατόπεδο αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι πάρα πολύ επικριτικό όσον αφορά κάνει αυτή η εταιρεία, αλλά και δεν βλέπω εγώ το λόγο για τον οποίο θα πρέπει να ήταν διαφορετικά τα πράγματα και εγώ διαρωτώ με κατά πόσον αυτή η επιτροπή ε, τι σκοπό εξυπηρετεί. Μόνο για αυξάνει τα έξοδα και τα πάνε οι οποίε έχουν οι διοικητικέ και οι γραφειοκρατικέ εταιρείε. Κύριε Λίγκον πρώτο έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους ομιλητές όλους που τόνισαν ότι πραγματικά σε αυτές τις εποχές ε, οικονομικής κρίσης είναι σημαντικό να επενδύσουμε σε μεταφορές και υποδομές. Και γι' αυτό θα ήθελα να σε επιστήσω την προσοχή στο πρόγραμμα «Μάρκο Πόλο». τι θέλουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε Επιτροπή Μεταφορών να πετύχουμε, κοιτώντας τον προϋπολογισμό για το 2009 και για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2010, από τα 54 εκατομμύρια πέφτουμε στα 30 εκατομμύρια σε ό,τι αφορά τις πληρωμές. Μιλάμε για τεράστια ποσά μείωσης. Και το, η πρόταση του Συμβουλίου είναι ακόμα μεγαλύτερη μείωση. Ο σκοπός που είχαμε πάντα με το πρόγραμμα του Μάρκο Πόλο ποιος ήταν η προώθηση των πλωτών μεταφορών. Όχι μόνο των θαλάσσιων μεταφορών, αλλά και των εσωτερικών πλωτών μεταφορών. Και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα αυτό και για τις εσωτερικές πλωτές. Να τονίσουμε λοιπόν αρκετά αυτές τις ε, εσωτερικές πλωτέ μεταφορέ. Γι' αυτό λοιπόν και προτείνω στην τροπολογία μου να επικεντρωθούμε ακριβώ στον τομέα αυτών. Γιατί ακριβώ σήμερα που είναι τόσο μεγάλε οι δυσκολίε που αντιμετωπίζει ο κλάδο αυτό, είναι σημαντικό να τονίσουμε τι ε, μεταφορέ αυτέ. Γι' αυτό λοιπόν σα ζητώ να υποστηρίξετε το κείμενο το οποίο προσθέτω να υποστηρίξετε την ε, τροπολογία μου που προτείνω στο, το κείμενο που προτείνω στο 6416 και θα ήθελα να συζητήσουμε με τον συνάδελφο Κόλιτσεκ. Μήπως θα έπρεπε να περάσουμε σε μεγαλύτερη πρόκληση, να μην βάλουμε μόνο 3 εκατομμύρια και να επανέλθουμε δηλαδή στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά να κοιτάξουμε τι έλεγε ο προπολογισμό το 2009. Δηλαδή, να θέσουμε πιο φιλόδοξους στόχους. Είναι σημαντικό φυσικά να είμαστε εναρμονισμένοι και να συμφωνούμε ο ένας με τον άλλον, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε και προς την κατεύθυνση της τροπολογίας της κυρίας Γένσεν προκειμένου να διευκρινίσουμε και ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ελσάντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τον κύριο Κόριτσα για τη δουλειά που έκανε καλοκαιριάτικα κιόλα, χωρίς πολλά πολυτεχνική υποστήριξη και να ευχαριστήσω και την Καταματία που τον βοήθησε. Θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζω όσα υπόθηκαν μέχρι τώρα, την ανάκτηση, την επιστροφή δηλαδή των κονδυλίων στην αρχική φάση του σε περίοδο κρίσης μάλιστα και τις ε, τροπολογίες που υποβάλαμε όπως αναφέρθηκε, στόχο έχουμε στην αποκατάσταση των αρχικών ποσών. Η κυρία Τικάου και αυτή τονίζει την ανάγκη αποκατάσταση των αρχικών ποσών και στον τουρισμό και στις μεταφορές. Είναι αναγκαία τα ποσά εδώ για να μπορέσει η Επιτροπή να υλοποιήσει τις δράσεις που ζήτησε το Κοινοβούλιο. Θέλω να υπογραμμίσω επίσης ότι πιστεύω, αυτό είναι καλό να το υπενθυμίσουμε, ότι οι μεταφορές και οι υποδομές ξεχάστηκαν από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάκαμψης και το Κοινοβούλιο είναι που το υπενθύμησε, σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό και να πω επίσης ότι υπάρχουν δύο τροπολογίες του κυρίου Κράμερ που δεν είναι θετικές και οι 6440 που αν κατάλαβα καλά μειώνει τις δράσεις μόνο στο ε, δρόμο του πλαισίου χάλιβα αλλά εγώ θα ήθελα ε, άλλα προγράμματα όπως αυτό το πρόγραμμα Ευρωποδήλατο σε μια, εγώ πρόγραμμα μια χώρα όπου προσπαθούμε τώρα να περάσουμε την κουλτούρα του ποδηλάτου Καλό θα ήταν να μην, ξεχνο, να μην ξεχνούνται. Κάποιες λοιπόν δράσεις από αυτό το Eurovelo θα ήταν σκόπιμο να φτάσουν και στις χώρες αυτές. Διαφωνώ λοιπόν με τις εκθέσεις αυτές. Το άλλο, η άλλη τροπολογία, η 6404, ε, αφορά και πάλι υποθέτω τη δική του περιοχή και επειδή ακριβώ εκεί βρίσκονται αλλά ε, καθοδόν εξελίξεις, αλλά δεν μπορούμε το Κοινοβούλιο σε μια κρίσιμη στιγμή όπως τώρα να λέμε ότι είμαστε κατά τη σχεδίων που ε, αποτελούν ένα από τα 30 προγράμματα του ΕΣΕΝ και πραγματικά δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι αντίθετο, θα μπορεί το Κοινοβούλιο να είναι αντίθετο με το σχέδιο αυτό. Κακό μήνυμα είναι αυτό και πιστεύω ότι θα έπρεπε να το αλλάξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κόχλιτσεκ για την έκθεσή του. Εγώ υπέβαλα ορισμένε τροπολογίες. Αναφέρθηκε βέβαια και από άλλους συναδέλφους αυτό. Πιστεύω ότι οι περικοπές ε, του προπολογισμού για τις υποδομές στα πλαίσια των μεταφορών δεν αποτελούν αποδεκτή λύση. Πρέπει να μεταφέρουμε το μήνυμα αυτό σαφώς, πόσο μάλλον που σε λίγο θα μιλήσουμε, θα, θα, έχουμε, θα συνομιλούμε με μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών ε, βαρύνουν περισσότερο στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Κάποιες από τι τροπολογίε αφορούν στην κατασκευή ασφαλών χώρων στάθμευσης, ε, ένα σημαντικό θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέσαμε κάποιες προποθέσει για το ε, ε, έχουμε θέσει για τους οδηγούς μια σειρά προϋποθέσεων, ώρες οδήγησης, ασφάλειας κλπ. αλλά και πρέπει να υπάρχει και, ένας, ε, και μια ρύθμιση ε, για τους ασφαλείς χώρους στάθμευσης για αυτούς. Ε, μέχρι τώρα αυτό δεν ίσχυε, αφορούσε μόνο, μια, υπάρχει μια πιλωτική μελέτη για μια περιοχή στα σύνορα Ευρώπης, νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης με τη Ρωσία. αλλά αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Επίσης υπέβαλα μια τροπολογία για τους ε, τουριστικούς προορισμούς ε, για τους καλύτερους ε, τουριστικούς προορισμούς, το οποίο θα ήθελα να επαναφέρει. Ζήτησε επίσης να υπάρχουν νέοι πόροι για τις δράσεις που αφορούν τα δικαιώματα των επιβατών. Να τονίσω εδώ το εξής, ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών που λάβαμε από τους Ευρωπαίους πολίτες μέχρι τώρα αφορούν ακριβώς μεταφορε, θέματα μεταφορών. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό να το πούμε, μια και μιλάμε για τα δικαιώματα των ε, ε, επιβατών. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα για την ε, δορυφορική πλοήγηση. Συζητήθηκε το θέμα αυτό. Συμπερασματικά θέλω απλά να πω ότι οι υποδομέ στον τομέα των μεταφορών μπορούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να αναπτύξουν την Οικονομική και τουριστική δραστηριότητα. Ευχαριστώ. Κύριε Ντουιρόν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Γεια σας. Εγώ είμαι νέο μέλος και ένα πληρωτήμα διαιτικό. Και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω την εργασία που έκανε ο εισηγητής και οι συνάδελφοι για αυτό το μέρος του προπολογισμού και να πω τα καλά λόγια τα οποία είπαν και προηγουμένω οι συνάδελφοι όσον αφορά την επένδυση που θα πρέπει να γίνουν για τις υποδομές και για τις μεταφορές αλλά βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει και μια ζήτηση, μια συμμήτηση η οποία θα έχει σχέση με την οικοδόμηση, η δόμηση οτιδήποτε τσουλάει θα έλεγα ιδιαίτερα σε αυτήν την περίοδο της κρίσης και εγώ είμαι στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και θα είμαι πάρα πολύ προσεκτική όσον αφορά τα αιτήματα της δική μας εδώ Επιτροπής θα περνάνε από την την Επιτροπή Προπολογισμών και όσο μπορεί αυτό να εισακουστεί. Εμεί θα είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι επίση ε, όσον αφορά τη συνάντηση κορυφή τη Κοπενχάγη σε θέματα τα οποία άπτονται ημών και των μεταφορών, καθώ επίση και ο φάκελο Μάρκο Πόλο, Γκαλιλαίο, και γνώρισα πολύ καλά με την κυρία Ντεπαλάωση όταν ξεκινήσαμε, το, το, το στην Βέλγικη Προεδρία της ΕΕ νομίζω πως είναι ντοσιέ τα οποία μεταφράζουν πάρα πολύ καλά την ανάγκη για την εργαστούμε την τεχνολογία επί της τεχνολογίας αλλά η τεχνολογία δεν επιλύει όλα τα πρόβληματα χρειάζεται πολύ περισσότερο αλλαγή, μια συμπεριφορά των οικογενειών, των νοικοκυριών για να δώσουμε πραγματικά ένα σήμα εμεί, αυτή τη στιγμή στι παραμονέ τη Κοπενχάγη όσον αφορά τη μείωση η οποία θα πρέπει να γίνει σε αυτό το τομέα και ότι βεβαίω θα πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή όσον αφορά τι επενδύσει που γίνονται και ιδιαίτερα τα νοικοκυριά τα οποία θα πρέπει να συμπεριφέρονται με διαφορετικά ε, ε, στο μέλλον. Και εδώ συνάδω πραγματικά με τους πράσινους συναδέλφους μου εδώ σε αυτή την επιτροπή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο επόμενος αγορητής, έσχατος, της Γραντές Πασκουά. Τη Γραντές Πασκουά. Εκτός μικροφώνου. Can the interpreters hear anything from... Τώρα λειτουργεί. Ευχαριστώ. Έλεγα ότι θα ευχαριστώ τον εισηγητή που έκανε μια πολύ αποτελεσματική δουλειά καλοκαιριάτικα όπως είπαν και προηγουμένως, όπου εμείς είμαστε σε διακοπές. Διπλάς ευχαριστίες και ευχαριστώ και τις υπηρεσίε που τον βοήθησαν. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ικανοποιητικά αυτά που μας είπε ο συντονιστής μας, εν γέννη, να αναφερθώ σε δύο τροπολογίες που είχα υποβάλει την επιστροφή των πιστώσεων για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας. Δεν μπορούν τα κονδύλια αυτά να μειωθούν ενώ η υπηρεσία όπως γνωρίζουμε θα αποκτήσει νέες αρμοδιότητες πρώτα με βάση τον κανονισμό και αργότερα πραγματικά νέες αρμοδιότητες. Δεν χρειάζεται λοιπόν, δεν πρέπει να κάνουμε περικοπές εδώ. Δεύτερον, την αποκατάσταση του αρχικού ποσό των προγραμμάτων Γαλιλαίο. Αναφέρθηκε τον Γαλιλαίο, αλλά και το έγνος, το πρόγραμμα είναι πίσω στο παρελθόν. Εγώ είχα εκφράσει τη λύπη μου διότι από τα τρία προβλεπόμενα κέντρα ελεγχού το τρίτο που ήταν στην Ισπανία, που ανήκε στην, στην αρμοδιότητα της Ισπανίας, καθυστέρησε και θα επιβαρύνει τη χώρα. Τέλο πάντων, έτσι έγιναν τα πράγματα. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε την ταχύτητα ενό ρυθμού που είναι τόσο σημαντική. Ενό προγράμματο τόσο σημαντικού. Ξέρουμε ότι τα προγράμματα είναι προγράμματα χρηματοδότηση και από την Ένωση και από τα κράτη-μέλη, αλλά δεν μπορούμε να μειώσουμε το, τις πιστώσεις σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά και ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Τεσλέντεγκραντες Πασκουάλ. Ο κύριος Φιλίππη για την Επιτροπή. Πού είναι ο κύριος Φιλίπη, <coughs> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για τις προτάσεις να, αποκατασταθούν, να αποκατασταθούν τα αρχικά ποσά του προσχεδίου προπολογισμού. Σας ευχαριστούμε ωστόσο την προσοχή στα εξή. Συνολικά, οι τροπολογίες που υποβλήθηκαν έχουν στόχο στην αύξηση και των πιστώσεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών. Το Συμβούλιο, ωστόσο, στην πρώτη ανάγνωση περιέκοψε όχι μόνο τις πιστώσεις στον προϋπολογισμό, αλλά και κάποιες θέσεις. Άρα θα μειωθούν και τα ποσά αντίστοιχα. Στις προτάσεις, στις τροπολογίες που έχετε υποβάλει στην Επιτροπή, υπάρχουν, και το ευχαριστούμε, τροπολογίες που αποκαθιστούν πιστώσεις. Όχι ωστόσο θέσεις που έχουν περικοπεί από το Συμβούλιο. Ωστόσο, χωρίς την αύξηση των θέσεων, οι περισσότερες πιστώσεις που προβλέπονται στις τροπολογίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Θα ζητούσε λοιπόν η Επιτροπή από εσά να λάβετε και αυτή τη διάσταση υπόψη και να υποβάλλετε μια τροπολογία που θα αποκαθιστά τις θέσεις που περιεκόπησαν από το Συμβούλιο. Μάρκο Πόλο τώρα. Συμφωνούμε με την τροπολογία που έχει στόχο να αποκαταστήσει τις πιστώσεις που είχε προτείνει το προσχέδιο προπολογισμού. Δεν βλέπουμε ωστόσο κατά πόσο είναι αναγκαίο να αυξηθούν οι πιστώσεις πληρωμών πάνω από τα 30 εκατομμύρια που ήταν το ποσό που είχε προτείνει η Επιτροπή στο προσχέδιο προπολογισμού. Γιατί διότι η μείωση των πληρωμών, των πιστώσεων πληρωμών που περιέχεται στο προσχέδιο προπολογισμού είναι αποτέλεσμα μιας μείωσης των προσκλήσεων υποβολή προσφορών που είχαν ξεκινήσει το 2008 και που πρέπει να πληρωθούν κατά πάσα πιθανότητα το 2010. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα το 2010 θα υπάρχουν λιγότερε ανάγκε πιστώσεων πληρωμών για το 2010. Επίση, διότι οι αλλαγέ που έγιναν στον κανονισμό Μάρκο Πόλο στο πρόγραμμα και που θα εντεθούν σε ισχύ το 2010 μόνο, θα σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν πληρωμές πραγματικά την ίδια χρονιά. Θέλω να σας ε, ε, διαβεβαιώσω ότι ο, η περικοπή αυτή δεν έχει καμία σχέση με το... Δεν σημαίνει ότι μειώνονται τα λεφτά των σχεδίων. Υπάρχει αύξηση 2 εκατομμύρια στις υποχρεώσεις. Αυτό που πρότεινε η Επιτροπή είναι μείωση στις πιστώσεις, στις, στις πιστώσεις πληρωμών, διότι λαμβάνουμε υπόψη την, το, το, την κατάσταση των, ε, πληρωμών, των πιθανών πληρωμών μέσα στο 2010. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 64-24, συμφωνούμε βέβαια για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, έχουμε κάποιες επιφυλάξεις για, την, για τις ε, παρατηρήσεις που υπάρχουν, τις αλλαγές στην, παρατήρηση, στην αιτιολόγηση. Κάποια τα ανέφερε ο κ. Γκρός. Πιστεύουμε ότι κάποιες από τις δράσεις που προτείνονται είναι, δεν είναι επιλέξιμες ή δεν συμφωνούν με τον κανονισμό διευρωπαϊκών δικτύων ή τις οδηγίες. Αν θέλετε, μπορούμε να δώσουμε στη γραμματεία τις προτάσεις μας για τις αλλαγές στην 64-49 ασφάλεια μεταφορών ε, εμείς θεωρούμε ότι η αύξηση που προτείνεται στην τροπολογία δεν είναι αναγκαία και νομίζουμε ότι μπορεί να καλυφθεί η ανησυχία στο επόμενο χρηματοδοτικό έτος. Εμείς έχουμε μια μικρή αύξηση μόνο στις ε, πληρωμές και στις ε, υποχρεώσεις. Τώρα για το πιλωτικό πρόγραμμα ασφάλεια στα, στα διευρωπαϊκά δίκτυα 6431 θα προτιμούσαμε να υπάρχει μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των υφιστάμενων έργων αυτών που χρηματοδοτήθηκαν το 8 και το 9 πριν δοθούν νέες πιστώσεις στο αυτό το πρότυπο σχέδιο. 64-57. Πρόκειται για μια νέα γραμμή προπαρασκευαστική δράση για την διευκόλυνση της διασυνοριακής κυκλοφορία στα, εξωτερικά στα νοτιοανατολικά εξωτερικά σύνορα τη Ένωση. Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι η πρωτοβουλία το 2009 βελτίωσε την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης με τη Ρωσία. Αυτό όμως αποτελούσε συνέχεια μιας αξιολόγησης που έκανε μια ομάδα εργασίας και που είχε δημιουργηθεί στον διάλογο μεταφορών μεταξύ Ένωσης και Ρωσίας που εντόπισε συγκεκριμένες προτεραιότητες για να εξασφαλιστεί ένα επαρκές επίπεδο ασφάλειας και υγιεινής για τους οδηγούς και το εμπόρευμά τους. Επιπλέον η δημιουργία χώρων ε, ανάπαυσης για τους οδηγού υπάρχει ήδη ε, χρηματοδοτείται ήδη μέσω δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δωρεών, ε, οικονομικών ενισχύσεων και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Κατά που άποψη επιτοπίζει λοιπόν η 64-57 τροπολογία δεν χρειάζεται. Εν τέλει, 64-58 έγνωση και Γαλιλαίο. Η Επιτροπή έχει την άποψη ότι η αύξηση κατά 50 εκατομμύρια στις πληρωμές δεν είναι αναγκαίο εν ώψη της ε, ε, κατάστασης υλοποίησης του έργου. Όπως είπε και το Μάρκο Πόλο, και εδώ δεν πρόκειται, δεν, έχουμε, δεν υποστηρίζουμε αύξηση στις υποχρεώσεις, αλλά δεν έχουμε πρόβλημα με την αύξηση στις υποχρεώσεις, αλλά με την αύξηση στις πληρωμές, που θεωρούμε ότι δεν είναι αναγκαίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Βόιτσεκ. Αν θέλετε να Uh, uh, θα είμαι σύντομο. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Σε τέτοιε εποχέ κρίση θα πρέπει να λάβουμε θετικά μέτρα. Δεν θα πρέπει να αυξήσουμε την ε, γραφειοκρατία και θα πρέπει να επενδύσουμε στις υποδομές και μάλιστα να επενδύσουμε σωστά, όπως είπε η κυρία Λεχτεμπέργκερ. Νομίζω λοιπόν ότι συμφωνούμε ουσιαστικά. Απλά θα πρέπει να συζητήσουμε αυτά που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι και με την κυρία Βόρτμαν Κόλ θα πρέπει να κάτσουμε και μαζί με τον κύριο Φιλίππη για να συζητήσουμε την τροπολογία της κυρίας Βόρτμαν Κόλ και να προτείνουμε τον τρόπο που θα συνεχίσουμε και να περάσω στα τσεχικά Μια και έχω τη δυνατότητα να μιλήσω τη γλώσσα μου να συνοψίσω λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να χτενίσουμε κάπως τις τελευταίες μας προτάσεις και ελπίζω ότι αύριο θα είμαστε σε θέση να τις ψηφίσουμε και ελπίζω ότι και με την υποστήριξη των νέων συναδέλφων να καταφέρουμε να περάσουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Να σας υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία για την έκθεση αυτή θα λάβει η χώρα αύριο στις 9 και 10. Ωραία, λοιπόν, κλείνουμε και αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Το επόμενο θέμα είναι η ανταλλαγή απόψεων για τις προτεραιότητες της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Μετά από τη συζήτηση τον Ιούλιο, με την, το Γενικό Διευθυντή Ρόιτερ. Μα μου φαίνεται ότι είναι η σωστή στιγμή να συζητήσουμε στα πλαίσια της Επιτροπής τις προτεραιότητες στις οποίες επιθυμεί η Επιτροπή μας να εστιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προκειμένου να μιλήσουν και οι νέοι βουλευτές. Θα θυμάστε, συνάδελφοι, ότι κατά τις συζητήσεις με τον κύριο Ρόιτερ, πολλοί βουλευτές τόνισαν κάποια σημεία από τη χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων, τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης, που θα τον αναφέρουμε στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, η ενδεχόμενη εφαρμογή και θέση σε ισχύ της ε, συνθήκης της Λισαβόνας, αλλά και η εφαρμογή της νομοθεσίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των επιβατών. Τη σημασία της επικοινωνίας με τον πολίτη, αυτό ήταν πραγματικά ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Τονίστηκε και στις ευρωεκλογέ. Όλοι επιθυμούσαμε πιο μεγάλη επικοινωνία με τους πολίτες, η ασφάλεια στις αερομεταφορές και τα υγρά και η καταπολέμηση της αλλαγής ε, του κλίματος και η βιώσιμη εξέλιξη όλου του τομέα των μεταφορών. Ακόμα και θέματα πειρατείας στη θάλασσα. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Φαίνεται ότι εξαφανίζονται πλέον και πλοία. Νομίζω λοιπόν ότι είναι καλή χρονική στιγμή να ακούσουμε τους νέους βουλευτές. Να τους δώσουμε λίγο χρόνο να συζητήσουν τις προτεραιότητες αυτές. Για να δώσουμε, αν θέλετε, και μία ένδειξη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το τι θέλουν οι αιρετοί βουλευτές να απασχολήσει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον. Να τηρήσουμε ωστόσο το χρονοδιάγραμμα Και να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γκρός. Ναι, εσείς είστε υπεύθυνε. Μάλιστα. Κύριος Γκρός, λοιπόν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση για τις προτεραιότητες θα την επαναλάβουμε πολλές φορές στους επόμενους μήνες. Έγινε και η συζήτηση τον Ιούλιο. Έχουμε ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μία μικρή εισαγωγή για το Λευκή Βίβλο, την οποία αναμένουμε του χρόνου, το 2010. Και το εννοώ όταν λέω μικρή εισαγωγή. Και νομίζω και ελπίζω σήμερα η ανταλλαγή απόψεων να αποτυπώσει και τα προγράμματα των διαφόρων ομάδων για τα διάφορα θέματα. Διάφορα θα είναι σημαντικά θέματα σε ό,τι αφορά την ενέργεια και το περιβάλλον, το οποίο αφορά διάφορα είδη μεταφορών. Ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί τόσο στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πέρα από τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερο θέμα, θεωρώ, το θέμα, το θέμα της ασφάλειας. Αυτό που αναφέρθηκε ήδη περιλαμβάνεται στην ε, ασφάλεια, νέες τεχνολογίες για την έρευνα, για τα αυτοκίνητα και θα πρέπει στον τομέα αυτό να θέσουμε σαφές, ε, σαφείς γραμμές. Και τέλος, μία ιδέα την οποία θα μπορούσαμε να ξαναδοκιμάσουμε εδώ στην Επιτροπή αυτή. Οι μεταφορές σε σχέση με την οικονομία. Γιατί έχουμε πολλέ φορέ την αίσθηση ότι καλύτερα να είναι φτηνέ οι μεταφορέ και όχι ποιοτικά καλύτερα. Καλύτερα δηλαδή να μειωθεί το κόστο παρά η αξιοπιστία. Νομίζω ότι σε αυτό το τομέα πραγματικά θα πρέπει να θέσουμε το αποτύπωμά μας. Και αυτό δεν θα γίνει από μόνο του και αυτό λοιπόν επανέρχομαι στο αγαπημένο μας θέμα. Τι θα κάνει το Συμβούλιο. Νομίζω ότι ως Επιτροπή Μεταφορών θα πρέπει μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να θέσουμε το δικό μας αποτύπωμα. Το θέμα δεν είναι να γίνει η εφαρμογή και όπως γίνει Το θέμα είναι η αξιοπιστία της εργασίας μας, αλλά και να υπάρχει ένας συνολικός προγραμματισμός. Και το θέμα είναι ότι πολλέ φορέ θέματα που συζητιούνται εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο και υπογράφονται από το Συμβούλιο δεν εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη. Διαπιστώνουμε, για παράδειγμα, ότι ζητάμε, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το χρόνο ανάπαυσης ελέγχους 2 έως 3%. Κι όμως πολλά κράτη λένε ότι δεν έχουν ε, τους απαραίτητους πόρους για να δεξάγουν τους ε, ελέγχους αυτούς. Εμείς μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραίες προτάσεις. Αν όμως δεν υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος στα κράτη-μέλη, είτε στις οδικές μεταφορές, είτε στις αερομεταφορές, τι νόημα έχει. Νομίζω ότι αυτές οι προσεγγίσεις θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Μιλήσαμε και για τις ε, υπηρεσίες, τα πρακτορία. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες, κάποια προβλήματα με τις υπηρεσίες αυτές, γιατί υπάρχει η αίσθηση ότι χρηματοδοτούνται μόνο διοικητικές εργασίες. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα διοικητικά έξοδα θα πρέπει να υπαθούν σε άλλους τομείς και όχι στις μεταφορές, αλλά πιστεύω ότι οι υπηρεσίες αυτές θα έπρεπε να παρουσιάσουν ποια είναι η προστιθέμενη αξία του σε ευρωπαϊκό επίπεδο και νομίζω ότι στο σημείο αυτό υπάρχουν θεωρητικά θετικές προσεγγίσεις για το πού μπορούν να συνεισφέρουν τα κρατη Και τέλος θα ήθελα να πω και το εξής. Συνολικά, σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, αποφασίσαμε για τα δικαιώματα των επιβατών σε πολλούς τομείς. Αυτό θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα να δούμε πώς θα ακολουθήσει η εφαρμογή. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν συμβάσεις από 7 πλευρές για το πού πρέπει να διαβάσει τα δικαιώματα του επιβάτης Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη απλοποίησης. Αυτό απλά το θέτω ως ιδέα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, το περιβάλλον και την αποδοτικότητα. Όλα αυτά αποτελούν τομείς που άπτονται των μεταφορών και νομίζω ότι σε αυτό το θέμα θα πρέπει να θέσουμε νέες ιδέες για το μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντω, του επόμενου μήνε θα έχουμε πολλέ ευκαιρίε, πιστεύω, για να κάνουμε μια γενική συζήτηση. Κάναμε μια πρώτη συζήτηση πριν από τι καλοκαιρινέ διακοπέ. Και υπάρχει και πλέον ε, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, έχουμε και τη συζήτηση με τους νέους ε, επιτρόπους που θα διοργανωθούν και θα ακολουθήσει και η Λευκή Βίβλος του χρόνου. Όλα αυτά είναι πολύ χρονοβόρα, αλλά θα μας δώσουν και ευκαιρίες να σκεφτούμε καλά. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το όλο συγκείμενο, το όλο πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε σήμερα. Δηλαδή, ε, θα ακολουθήσει στα τέλη του έτους η συνάντηση για το κλίμα της Κοπενχάγης. Δεν νομίζω ότι μπορούμε λοιπόν να απομονώσουμε τις εργασίες μας από αυτό το πλαίσιο. Θα πρέπει να συνδεθούμε και με τη συζήτηση αυτή. Αφετέρου έχουμε και την οικονομική κρίση. Για την ομάδα μου υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Καταρχάς, το συζητήσαμε ήδη άλλωστε, και σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό. Είναι λοιπόν σαφέ ότι οι επενδύσει θα πρέπει να αυξηθούν, όχι να μειωθούν οι επενδύσει στι καλύτερες και περισσότερες υποδομές. Αυτό θα αποτελέσει μέρος της αντιμετώπισης της κρίσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί και η μελλοντική ανάπτυξη. Δεν θα πρέπει βέβαια αποκλειστικά να έχουμε κατά νου περισσότερα κονδύλια. Νομίζω ότι η έκθεση η περσινή για το πώς έχει η κατάσταση για τον Μάρκο Πόλο κατέδειξε ότι σε ό,τι αφορά θέματα γραφειοκρατίας και διαδικαστικά θέματα μπορεί να σημειωθεί πρόοδος προκειμένου να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν καλύτερα οι ήδη φυστάμενοι πόροι. Άρα, σημειώθηκε πρόοδος, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω η κατάσταση. Κάτι άλλο. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε πιο εθελούσια, αν θέλετε, διοίκηση για να πετύχουμε πιο, βιώσιμες, ε, πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς. Μιλάμε για τα προγράμματα ΣΕΖΑΡ, για την τεχνολογία, για την εισαγωγή προτύπων σε ό,τι αφορά τα οχήματα και για την λιγότερο ακριβή εφαρμογή νέων προτύπων. Ένα τρίο, τρίτο κεφάλαιο είναι όλα όσα άπτονται του χρήστη των μεταφορών. Μίλησε ο συνάδελφος Γκρός για τα δικαιώματα του επιβάτη. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια κάναμε κάποια βήματα προς την ε, σωστή πλευρά. Το πρόβλημα όμως είναι ότι υπάρχουν κενά στην εφαρμογή. Νομίζω ότι από κοινού με την Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να κάτσουμε να κοιτάξουμε και να δούμε πού χρειάζονται πιο ε, αυστηρά μέτρα για να είναι σωστή η εφαρμογή. Για παράδειγμα, μια αεροπορική εταιρεία η Sky Europe, και φαίνεται ότι δεν έχουμε ακόμα ταμείο εγγύησεων για τέτοιες ε, ε, αεροπορικές εταιρείες σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά ταξίδια. Δηλαδή υπάρχει τέτοιο ταμείο για ταξίδια αναψυχής μέσω γραφείων, αλλά όχι για τις αεροπορικές εταιρείε. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Κάτι άλλο. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την ε, ασφάλεια στις μεταφορές θα πρέπει να σημειώσουμε καινούργια πρόοδο. Γιατί κάθε χρόνο 40.000 είναι νεκροί στα ευρωπαϊκά δίκτυα. Έχει μειωθεί αυτός ο αριθμός βέβαια σε σχέση με πριν από κάποια χρόνια. Αλλά παρόλα αυτά είναι απαράδεκτο, απαράδεκτα υψηλά, ο υψηλός αριθμός αυτός. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να, θετου, να θεθούν νέοι στόχοι αυτό και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, αυτό πιο εσωτερικό θέμα αν θέλετε για την Επιτροπή μας. Θα πρέπει να κοιτάξουμε την επιτροπολογία με έλεγχο και θα πρέπει να συνεχίσουμε να αντιδραματίζουμε το ρόλο μας ως Κοινοβούλιο όχι μόνο κατά την κατάρτιση της νομοθεσίας αλλά και κατά την ε, τροποποίηση αν θέλετε μικρών στοιχείων, λεπτομεριών. Θα πρέπει λοιπόν να παίξουμε το ρόλο μας ως θεματοφύλακας και στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λίχτεμπέργκερ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες θα ήθελα να συμφωνήσω με τον συνάδελφο Γκρός. Διαπιστώνουμε στο Συμβούλιο ότι η εφαρμογή στα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα θέματα ελέγχου. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η εφαρμογή αυτή είναι τόσο καθυστερημένη που πραγματικά καθίσταται αντιπαραγωγική. Νομίζω ότι για μας ε, στην Επιτροπή Μεταφορών είναι κατεπίγουσα ανάγκη να εξετάσουμε τα θέματα αυτά. Το κάνει άλλωστε και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων να δούμε λοιπόν πού είναι τα ελλείμματα σε ό,τι αφορά τη μεταφορά, την εφαρμογή της νομοθεσίας, πού υπάρχουν τα μεγαλύτερα κενά και τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς για να βελτιωθεί η κατάσταση. Κοιτώντας λοιπόν την κατάσταση σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τον ευρωπαϊκό έλεγχο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σε ό,τι αφορά τους χρόνους ανάπαυσης. Πραγματικά μου να βάλω τα κλάματα. όταν βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη να δράσουμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται. Θα πρέπει λοιπόν να ρωτηθούμε, έχει νόημα η ευρωπαϊκή ρύθμιση. Αν λοιπόν καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ναι, υπάρχει δυνατότητα να ρυθμιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το θέμα και τελικά τα κράτη-μέλη έρχονται και δεν εφαρμόζουν, δεν μεταφέρουν την νομοθεσία, ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με το θέμα αυτό. Γιατί υπάρχουν... Γιατί μάλλον σε αυτό οφείλονται προβλήματα όπως η αύξηση των εκπομπών. Για παράδειγμα, να σας υπενθυμίσω ότι οι μεταφορές σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ευρώπη ιδιαίτερα είναι ο τομέας με, τις μεγαλύτερες, με τη μεγαλύτερη αύξηση των εκπομπών. Με άλλα λόγια δηλαδή, η ίδια μηχανία. Ε, οι πολίτες επενδύουν χρήματα για να μειώσουν τις εκπομπές τους. Και έτσι αυξάνεται το κόστος των επενδύσεων. Και τελικά τι συμβαίνει, όλες αυτές ε, οι προσπάθειες μείωσης αντισταθμίζονται από την αύξηση των εκπομπών στις μεταφορές. Ε, αυτή την κατάσταση δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχιστεί Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα πρέπει να το συζητήσουμε. Λοιπόν, για το πώς μπορούν να μειωθούν οι εκπομπές. Για παράδειγμα, συστήματα διαχείρισης της ζήτησης σε ό,τι αφορά το Single Sky, για παράδειγμα. Ποια είναι τα κρατη που δεν συνεργάζονται και σε ό,τι αφορά το εξωτερικό κόστος στις μεταφορές, να συμπεριληφθούν και τα ε, αυτοκίνητα, που και πάλι τα κρατη είναι αυτά που μπλοκάρουν την ε, κατάσταση. Για το θέμα των υπηρεσιών τώρα και το κατά πόσο είναι απαραίτητες ή κατά πόσο μπορούμε και να τις αποφύγουμε, όπως λένε οι Βρετανοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε και με, κριτική, με κριτικό βλέμμα. Τα κράτη-μέλη μπορούν να εξοικονομήσουν πολύ προσωπικό με τέτοιες λύσεις. Αλλά όταν υπάρχουν προβλήματα, αυτά δεν οφείλονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο, οφείλονται στο κράτη-μέλη σε διάφορες νομικές καταστάσεις. Ίσως να πιστεύουν και κάποια κράτη-μέλη ότι είναι τα μόνα που μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση. Εδώ λοιπόν πραγματικά θα πρέπει να εξετάσουμε με προσοχή τι γίνεται. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδεροδρόμων, το ότι είναι απολύτως απαραίτητη, νομίζω κατέστη σαφές μετά από το καλοκαίρι. ταξίδεψα με το τρένο και είδα ποια είναι τα ελλείμματα. Ή βλέπουμε με σαφήνεια ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σιδηροδρομοί. Να υπενθυμίσω στα μέλη ότι όταν σηκώνω αυτό το σφυράκι δεν είναι για να σα απειλήσω, αλλά θα πρέπει να περατώνετε. Αυτό είναι ο λόγο για το οποίο σηκώνω το σφυράκι. Ο κύριο Στερξ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι ακούστηκαν τα πιο πολλά στοιχεία. Το πιο σημαντικό ή ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι η βιωσιμότητα ασφαλώς, όπου δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ της οικονομίας και των μεταφορών, της κινητικότητας. Βλέποντας λοιπόν την κρίση που περνάμε σήμερα και τι, ποιος είναι ο αντίκτυπος για τις ε, ροές μεταφορών, βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι δραματική σήμερα έχουν περιοριστεί οι μεταφορές. Αυτό διαπιστώνουμε και θα πρέπει να φροντίσουμε τη βιωσιμότητα των ε, ροών μεταφορών. Γιατί αν θα βελτιωθούν οι μεταφορές δεν θα ανακάμψει ποτέ και η οικονομία. Οι ροές αυτές θα αυξηθούν κατά πάσα πιθανότητα τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να εγγυηθούμε ότι θα είναι αποδοτικές και αποτελεσματικές. Γι' αυτό λοιπόν τίθεται θέμα προϋπολογισμού στις υποδομές, στα διευρωπαϊκά δίκτυα, αλλά θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό μια δεύτερη πτυχή. Είναι η σχέση με την ενιαία ιστορική αγορά. Μιλάμε για τον έλεγχο των αερομεταφορών, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα όπως είπε η κυρία Λίχτενμπέργκερ, το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη ουσιαστικά δεν θέλουν να υπάρχει ευρωπαϊκή ρύθμιση. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των μεταφορών και θα πρέπει στο σημείο αυτό να πούμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και ε, μπλέκονται πάρα πολλά θέματα, φορολογικά, κοινωνικά, αλλά να μην ξεχνάμε ποιος είναι ο στόχος μας για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Ο κύριος Αλκαντράουι επίσης έδειξε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε την ασφάλεια των μεταφορών. Γιατί αυτό αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το τονίσουμε ως Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο. Στο σημείο αυτό πιστεύω ότι είμαστε πολύ αργοί και καθόλου αποτελεσματικοί. Είτε με οδηγίε, είτε με καλύτερες πρακτικές. Να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε δραστικά τα αποτελέσματα αυτά. Νομίζω ότι θα τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά και τους επόμενους μήνες. Σίγουρα και σε ό,τι αφορά τα θέματα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών θα έχουμε σίγουρα πολλή δουλειά. Και οι προτεραιότητες αυτές θα ανακύψουν από μόνες τους. Και σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της Λευκής Βίβλου θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πάλι τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Ντιβέρακ, παρακαλώ, έχει το λόγο. Κυρία Ντιβέρακ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ ότι γίνεται αυτή η συζήτηση όσον αφορά τι προτεραιότητε, για τις μεταφορές τα επόμενα χρόνια διότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να υιοθετήσουμε πάρα πολλά κείμενα τα οποία είναι σημαντικά. Υπάρχουν μεγάλα project τα οποία θα πρέπει να εκκρεμούν και θα πρέπει να γίνουν και θυμάμαι την οδηγία Μομπινιέ και όσον αφορά την ασφάλεια την αεροπορική και αύριο θα πρέπει να ρωτήσουμε τη Σουηδική Προεδρία για τις δραστηριότητες τις οποίες θα πρέπει αυτή τη στιγμή να αναπτύξει για να προχωρήσουν αυτά τα κείμενα. Θα ήθελα επίσης να μοιραστώ μια σκέψη μου μαζί σας. Η Επιτροπή Λοιπόν συναρμόδιο είναι όσον αφορά τα θέματα της μετα, μετα, μεταρρύθμισης της αεροπορικής αερομετρικής ε, της αλλά όχι το τεχνικό μέλος. Θα πρέπει λοιπόν θα πρέπει να παρακολουθήσουμε εκ του τσίνιγκης τα θέματα εκείνα τα οποία άπτονται όσον αφορά το τεχνικό μέρος αυτού αυτό το θέμα, να έχουμε μια κρόαση, ένα hearing, επίσης να έχουμε πραγματικά τους εκπροσώπους της εταιρεία Σεζάρ, οι οποίοι θα μπορούν να έρθουν εδώ πέρα και να με παρακολουθήσουν τι θέλει να πει αυτό το θέμα. Πιστεύω το Σεζάρι είναι ένας παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός όσον αφορά την ανάπτυξη και παρακολουθεί το Γαλιλαίο και η Γαλιλαίο μας έχει δείξει ότι οι επιχειρήσεις που άπτονται αυτή ε, του project θα έχουν την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να σας πω το εξή για τις προτεραιότητες. Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό ενιαίο θαλάσσιο χώρο. Φέτος το καλοκαίρι ωστόσο η πειρατεία ήταν αυτή που ε, κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα και αντιμετωπίσαμε ένα, ένα δυσάρεστο, μια σειρά δυσάρεστων ε, γεγονότων. Πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να μην μείνει το ζήτημα της πειρατείας μόνο σαν ένα ζήτημα άμυνας, αλλά και σε ένα ζήτημα μεταφορών. Θα έπρεπε λοιπόν να ακούσουμε τους εμπλεκόμενους στον τομέα για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να αντιμετωπίσουμε το θέμα της πειρατείας από την οπτική των μεταφορών. Κατόπιν, στην ασφάλεια των εναέριων μεταφορών είναι σημαντικό η Επιτροπή και επανέρχομαι και στο θέμα της επικοινωνίας με τους πολίτες την ανάγκη να περνάμε σε αυτούς τα νέα και τις πληροφορίες από τις ε, διάφορες αεροπορικές εταιρείες. Να μπορούμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουμε το θέμα όχι της αγοράς των υπηρεσιών, γιατί θα υπάρξουν τεράστια προβλήματα, αλλά κυρίως τουλάχιστον να πάμε παραπέρα από τα απλά δικαιώματα των ε, επιβατών σε ένα τομέα ποιότητας των υπηρεσιών, για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια πραγματική συζήτηση για την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. Επίσης, να αυξήσουμε τη συζήτηση για την κινητικότητα στις πόλεις. Ένα θέμα κοντά στον πολίτη και αυτό που θα έπρεπε να το ανακτήσουμε, ιδίως από επιμελητιακή οπτική γωνία, ε, με διαδρόμους, ε, με ποδηλατόδρομους, με μεγαλύτερη πεζοδρόμηση, να μιλήσουμε και για την ε, οδική ασφάλεια. Άκουσα για, να γίνεται λόγος πάλι για τις καλές πρακτικές στο Κοινοβούλιο. Υπάρχουν δύο εκκρεμή ζητήματα για την ε, οδική ασφάλεια. Ε, δεκαετίες ζούμε με καλές, με τις βέλτιστες πρακτικές που δεν λειτουργούν. Το θέμα του ορίου ταχύτητας είναι ένα βασικό το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Το ξαναφέρνω το συζήτηση, ξέρω ότι είναι αμφιλεγόμενο θέμα, αλλά τουλάχιστον να υπάρξει μία συμφωνία για το τι μπορεί να κυρωθεί, να, να τιμωρηθεί εφόσον είναι παράνομο οπουδήποτε. Θα μπορούσαμε να αναθεωρήσουμε τους στόχους του 2010 και να δώσουμε ένα σημαντικό μήνυμα, συμφωνώ με τον κύριο Αλκατράουη. Τέλος, τουρισμός. Το γεγονός ότι Θέλαμε να υπάρξει νομική βάση όταν, ε, αν εγκρινόταν το Σύνταγμα, τώρα αυτό μπλόκαρε, αλλά ε, πάλι όποτε προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του τουρισμού, μπλοκάρουμε σε αυτό το θέμα. Άλλοι έξι ομιλητέ υπάρχουν. Λέω θα παρακαλούσα του συναδέλφου να είναι όσο πιο σύντομα γίνεται. Κύρια Φώστερ πρώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ε, πολλοί συναδελφοί μέχρι αυτή τη στιγμή κάνω σχόλια πάρα πολλά όσον αφορά τη μεταφορά βεβαίω, αλλά δούμε αυτή τη στιγμή μιλάμε για προτεραιότητε. Έχει αυτό το σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα αν δω πραγματικά τα θέματα εκείνα τα οποία μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ είναι βεβαίως οι ενέργειες μεταφοράς. Ένα από την πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να μην έχουμε έναν υπερκανονισμό ο οποίο θα πρέπει διότι έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια του προπολογισμού ότι όλες οι οικονομίες περνάνε δύσκολες περιόδους και αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο πρέπει να ξέρουμε πραγματικά πού πάει τα χρήματα, πού πάνε τα χρήματα, συγγνώμη, και οι δικέ μα κυβερνήσει επίση, Ξέρετε, ξέρετε οι αερομεταφορές έχουν αυτή τη στιγμή κέρδη και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και βεβαίω υπάρχουν τεράστια κόστη αυτή τη στιγμή. Ο κ. Ντεβέιρα ανέφερε ε, και από την, ε, θα έρθει αύριο κάποιος ο οποίο θα μας δει ότι υπάρχουν πραγματικά υπάρχουν χρήματα τα οποία έρχονται προς την αερομεταφορές από τις εθνικές και ξέρετε αυτά τα θέματα είναι βεβαίως θέματα εθνικού προπολογισμού. Έτσι λοιπόν όταν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά τα θέματα ακουπής θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το εξή. ότι αυτή η επιτροπή είναι αυτή ε, πρέπει να δούμε τη βιομηχανική πλευρά αυτή τη στιγμή. Ξέρετε ότι υπάρχουν βιοτεχνίες, υπάρχουν πάρα πολύ εξειδικευμένα και ξέρετε υπάρχουν βιομηχανίες οι οποίες εργάζονται για αυτό το τομέα πολύ συγκεκριμένα και θα πρέπει είναι πραγματικά θα είναι οι επιπτώσεις θα έχουν γιατί αυτά θα πρέπει να απολυθούν. Θα πρέπει να το δούμε σφαιρικά λοιπόν το όλο θέμα. Τέλος θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να τα λάβει όλα αυτά υπόψη και θα έχουμε μια συζήτηση σημαντική και επικοδομητική όσον αφορά τη μεταφορά επιπτώσεις ε, επί του περιβάλλοντος επίσης να ληφθούν υπόψη και περέντος θα πω ότι δεν είναι μόνο η αεροβιομηχανία αλλά θα πρέπει να δούμε και τις θαλάσσιες μεταφορές και αυτός είναι τεράστιος τομέας και θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και θέτω εγώ αυτή την επιφύλαξη και ότι σε επόμενου μήνε θα έχουμε μια ει βάθο συζήτηση, ανδελεχή συζήτηση με την προσεχή τη δέωση που πρέπει να, να υπάρξει για αυτό το θέμα. Κύριε Βαντάλεν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μίλησαν διάφοροι συνάδελφοι για το θέμα της εφαρμογής και του ελέγχου, το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Θα ήθελα να προσθέσω ένα στοιχείο, ωστόσο, στη συζήτηση αυτή. Η Ειλικρινή έλεγχη και εφαρμογή. Να είμαστε δίκαιοι, γιατί πολλοί κλάδοι αναφέρουν ότι κάποιες εθνικότητες σε κάποιες χώρες αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από την ντόπιοι. Άρα θεωρώ ότι είναι σημαντικό όταν μιλάμε για εφαρμογή και έλεγχο να γίνονται με δίκαιο τρόπο όλα αυτά. Ένα δεύτερο θέμα είναι και η ασφάλεια το οποίο δικαίως ανέφεραν οι συνάδελφοι, να τονίσω στο πλαίσιο αυτό την πτυχή της επικοινωνία. Θα πρέπει με σωστό τρόπο να γίνεται η επικοινωνία. Και να τονίσω για παράδειγμα τον κλάδο των πλωτών ιστορικών μεταφορών, όπου χρησιμοποιούνται πολλές γλώσσες, για παράδειγμα η γλώσσα του πλοίου. Αλλά δεν υπάρχει ουσιαστικά μία κοινή γλώσσα και ξέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις κάθε χρόνο ε, υπάρχουν πολλά ατυχήματα επειδή δεν υπάρχει μια κοινή γλώσσα. Για παράδειγμα ένα πλοίο μιλάει γαλλικά, ένα άλλο πλοίο μιλάει γερμανικά. Και έτσι προκύπτουν προβλήματα. Άρα θα ήθελα να τονίσω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στις εσωτερικές πλητές μεταφορές να μην ξεχνάμε το στοιχείο της γλώσσας. Κάτι άλλο που είπε η κυρία Λίχτενμπέργκερ, το θέμα του κλίματος. Όντω ο μέσο των μεταφορών είναι ένα από του τομεί που προκαλεί τη μεγαλύτερη ρήπανση στην Ευρώπη. Πιο πολύ ρήπανση και από τη βιομηχανία. Ωστόσο υπάρχουν μεγάλες προοπτικές και θα πρέπει κυρίως να επικεντρωθούμε στην μείωση του νόξ των οξυδίων του αζότου, γιατί πολλές φορές εστιαζόμαστε υπερβολικά στο διοξίδιο του άνθρακα. Νομίζω ότι ε, αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Τέλος, είμαστε όλοι πολιτικοί και είμαστε σε διοικητικές ε, θέσεις και πολλές φορές μας αρέσει να καταρτίζουμε υπερβολικά πολλούς κανόνες αν θέλετε για να βελτιώσουμε τον κόσμο μας αλλά θα ήθελα να σας ε, καλέσω να είμαστε και να κοιτάμε με κριτικό ε, βλέμμα και τις ε, δράσεις μας, να δούμε μήπως ε, δεν χρειάζονται τόσοι πολλοί κανονισμοί, τόσο πολλή ρύθμιση. Θα πρέπει πραγματικά να εξετάσουμε σε κάθε περίπτωση αν υπάρχει το θέμα η αξία σε μια καινούργια απόφαση. Να είμαστε λοιπόν, να ασκούμε αυτοκριτική και να πατάμε και λίγο φρένο κατά καιρού. Θα πατήσω λοιπόν και εγώ φρένο. Πρόεδρε, γιατί βλέπω ότι σηκώνει το σφυρί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, παρακαλώ, πρέπει να με παρακαλώ. Δεν είπε το όνομα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα σημαντικό θέμα για τον, τη μακροπρόθεσμη περίοδο, γιατί άκουσα για τη Λευκή Βίβλο, για τη διάσκεψη της, Κο, της Κοπενχάς και Έχουμε και μπροστά μας και μια κρίση που θα επηρεάσει και τον τουρισμό και τις μεταφορές με πολύ έντονο τρόπο. Άρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προλάβουμε αυτό το μακροπρόθεσμο πλαίσιο που φαίνεται ακόμα πιο μεγάλο, πιο μακρύ τώρα και να δώσουμε άμεσα και αμέσως απαντήσεις. Τα στοιχεία που μας προτείνουν τα δημοσιονομικά όργανα είναι πολύ περιορισμένα σε σχέση με τις ε, υποχρεώσεις που υπάρχουν. Σε ό,τι αφορά την, τον έλεγχο της ασφάλειας, τις δημόσιες επενδύσεις, ε, πέραν αυτών θα ήθελα να ακούσω και για μια ε, κουλτούρα των ΣΔΙΤ, της σύμπραξης δημοσίων και ιδιωτικών πόρων, ούτως ώστε να προχωρήσουν ταχύτερα κάποια έργα από την συνηθή και από τις Δυνατότητε που προσφέρει οικονομική, κρατική οικονομική ενίσχυση. Θα έπρεπε λοιπόν να περάσουμε μια κουλτούρα και για το Κοινοβούλιο και για την Κομισιόν, καινούργια κουλτούρα, περνώντας από την δημιουργία μέσω του ιδιωτικού τομέα ή από την, την σύσταση ενός μεγάλου ευρωπαϊκού ε, κρατικού ενδεχόμενα ε, ταμείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την κάλυψη των αναγκών των μεταφορών και του τουρισμού ίσως φροντίζοντας ούτως ώστε στο ταμείο αυτό να μπορούν να μετάσχουν ιδιώτες και ανεξάρτητα και με αυτόνομο τρόπο και να επιτρέψουμε έτσι κάποια έργα να έχουν ένα ταχύ, ταχύτερη υλοποίηση σε ένα μέλλον εγκύτερο δημιουργώντας και δίνοντας σε κίνηση μια οικονομία που πάσχει παντού. Αυτή η κουλτούρα λοιπόν ε, λειτουργίες μέσω των συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να αναζητήσει την βελτίωση της δημόσιας συνδρομής του τομέα της ασφάλειας με την συνεισφορά του ιδιωτικού. Αυτό ήθελα να πω για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε την πορεία αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος ο νόμος της ανισόμετρης οικονομικής ανάπτυξης και ότι το γεγονός αυτή την περίοδο διανύουμε οικονομική κρίση, βαθιά οικονομική κρίση, θέτουν με μεγαλύτερη πίεση διαφορετικές προτεραιότητες και στα 27 κράτη-μέλη. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πραγματικά με τον α ή τον β τρόπο εκφράστηκε και από προηγούμενους ομιλητές. Πριν από λίγο συζητούσαμε σε ό,τι αφορά το σχέδιο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ό,τι αφορά τον τομέα ευθύνης της Επιτροπής Μεταφορών. Είναι πράγματι απογοητευτικό ότι δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση δαπανών το 2010 για συγκεκριμένα έργα όπως ο άξονας πολλαπλών μέσων μεταφοράς Ισπανίας-Πορτογαλίας-Ευρώπης για την οδική πρόσβαση πολλαπλών μέσων μεταφοράς Ιρλανδίας Μπενελούκ, για την κύρια σιδηροδρομική γραμμή Δυτικής Ακτής, για τους θαλάσσιους αυτοκινητόδρομους και άλλα σοβαρά έργα που πραγματικά έχει ανάγκη η Ευρώπη και οι λαοί της. Είναι γεγονός πραγματικά ότι είναι μεγάλα σοβαρά τα προβλήματα Νομίζω ότι δεν υπάρχει διαφορετική άποψη, ανεξάρτητα από ποια αφετηρία ξεκινάει κάποιος, ότι οι μεταφορές συνολικά είναι στρατηγική σημασίας τομέας σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Είναι γνωστά τα στοιχεία, θα ήταν πλεονασμός να τα αναφέρω. Τι θέλω να επισημάνω. Κατά καιρούς παίρνονται νομοθετικές ρυθμίσεις όπου η πορεία τους σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματά τους δεν ελέγχονται από τις επιτροπές, δεν ελέγχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να φέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα και να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Ενώ ήταν υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει έκθεση, την πέμπτη έκθεση, για τις εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές, από το 2004 διανύουμε το 2009, έχει διαμορφώσει μια έκθεση για τα συμπεράσματα μέχρι το 2005 και με καθυστέρηση 5 ετών, 6, θα έρθει να συζητήσει για αποτελέσματα τα οποία παράθηκαν μια προηγούμενη πενταετία. Τελειώνοντας θέλω να πω το εξή. Εκεί που πρέπει να εστιάσουμε και από την πλευρά μας ό,τι μας αφορά σαν ομάδα, σαν γκουε θα προσπαθήσουμε να φέρουμε στο τραπέζι των συζητήσεων στην Επιτροπή μας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι τα προβλήματα που αφορούν τους εργαζόμενους τόσο μισθολογικά εργασιακά αλλά και στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Κύριε Σαούτζιας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δέχομαι την πρότασή σας να μιλήσω για τις μεταφορές ως συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τα συγκεκριμένα προβλήματα των πολιτών και που αφορούν δικαιώματα στην κινητικότητα, στην κοινωνική ένταξη και στην οικονομική ένταξη. Εξίσου συγκεκριμένα θέλω να σας πω ότι όντως εγώ όπως και άλλοι εκπροσωπούμε ολόκληρη την Ευρώπη, ωστόσο δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και επενθυμίζω κάτι τέτοιο ότι είμαι νησιώτης όπως και εσείς πρόεδρε. Είμαι κατάγομαι από τη Σαρδινία που μαζί με τη Σικελία είναι οι δύο μεγάλα, τα δύο μεγάλα νησιά της Μεσογείου. Μετά το νησί του Προέδρου βέβαια, η Σαρδινία είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σικελία και η Σαρδινία, 7 εκατομμύρια κάτοικοι μαζί, είναι δύο περιφέρειες της Ευρώπης όπου δεν υπάρχει ούτε ένας αυτοκινητόδρομος. Στη Σαρδινία με 1,5 εκατομμύριο κατοίκους δεν έχουμε σύνδεση με το εθνικό και ευρωπαϊκό συνδρομικό δίκτυο. Η παρέμβασή μου λοιπόν ήθελε ακριβώς να αναδείξει ένα θέμα που θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στην επόμενη λευκή βίβλο μεταφορών, να δώσει την προτεραιότητα της απομόνωσης που αντιμετωπίζουν διάφορες περιοχές στην Ευρώπη. Και για να αναφέρω το γεγονός ότι στις περιφέρειες εκείνες τα πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής πολιτικής μετατρέπονται σε μειονεκτήματα, διότι οι καταστάσεις εκείνες τις οικονομίες με, την οποία, με τις οποίες διαφυλάσσεται, ε, εξασφαλίζεται συνδεδομική μεταφορά ή μείωση του κόστους στο περιβάλλον, στην ασφάλεια, στις ανθρώπινες, στην ανθρώπινη ζωή γίνεται υπερβολικά υψηλό. Κλείνω. Αν θέλουμε να περάσουμε στους πολίτες μας, στους Ευρωπαίους πολίτες, μια εικόνα Ευρώπης ευκαιριών και όχι μόνο Ευρώπης δεσμών, δεν πρέπει να κοφεύουμε στα αιτήματα των νησιωτών, Πρόεδρε. Well, thank you, Mr. Ευχαριστώ πάρα βεβαίως έχω αυτή τη στιγμή, επειδή έχω πάει σε διάφορα μέρη της Αρτινίας μπορώ να επιβεβαιώσω ότι πραγματικά είναι καταπληκτικό. Ο επόμενος παρακαλώ. Νομίζω πως πραγματικά πρόεδρο υπάρχουν θέματα τα οποία θέματα τα οποία τέθησαν είναι αυτή τη στιγμή η ασφάλεια. Ξέρετε ότι από το 2003 υπήρχε ένα σύστημα το οποίο έχει εισήχθη αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να ισχύει το 2006. Υπάρχει ένα μικρό μηχάνημα το οποίο αυτή τη στιγμή και μπορεί να εξασφαλίσει αυτή τη στιγμή όλου του παράγοντε εκείνου που έχουν σχέση με την άσφυνα, να την ασφάλει και να αποφύγει τα ατυχήματα. Και μπορεί αυτό το πράγμα να σημαίνει όσον αφορά τα ατυχήματα με τα αυτοκίνητα και κατα... πάρα πολύ πραγματικά ότι αυτή τη στιγμή ήρθε ο καιρός να σώζουμε τις ζωές αυτή τη στιγμή. 21 χώρες έχουν εισάγει αυτό το σχέδιο, αλλά έξι δεν το έχουν κάνει. Και η δική μου χώρα, η Ιρλανδία, είναι μέσα σε έξι. Πιστεύω λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό το μηχάνημα είναι τόσο αποτελεσματικό, τόσο αποδοτικό αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να υπάρξει μια οδηγία η οποία θα είναι υποχρεωτική για όλε τι χώρε τη περιλαμβανομένε και τη δική μα, για να υπάρξει αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει και το οποίο αποφεύγει τα ατυχήματα και βεβαίω κατά αυτόν τον τρόπο πραγματικά θα αποφύγουν πάρα πολλά ατυχήματα στο μέλλον. πάρα πολύ ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η ευκαιρία αυτή τη στιγμή στα μέλη να έχουμε μια συζήτηση αυτή τη στιγμή όσον αφορά μια αρχική συζήτηση όσον αφορά τις μεταφορές και, αυτό το, και τις προτεραιότητες που θα πρέπει έρθουν για τα επόμενα πέντε χρόνια της θητείας μας και ιδιαίτερα αυτή την παρουσίαση που μας έχει γίνει και φαίνεται πως υπήρξε πάρα πολύ επιτυχημένη αυτή και όταν δούμε το μακρύ κατάλογο των ομιλητών υπάρχουν άτομα τα οποία θέλουν να συμμετέσχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το οποίο χρειάζομαι χρειάζεται να δύο είναι ότι οι συντονιστές φίλοι μου ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό τον κατάλογο των ομιλητών συναδέλφων οι οποίοι και να δουν πραγματικά ποια είναι η θέση της Επιτροπής αυτής της Κομισιόν του Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα όταν έχουμε αυτή τη στιγμή με μια πρόταση της Κομισιόν για το 2010. Είναι λοιπόν αξίζει τον κόπο αυτή, αυτή η εργασία που πρόκειται να γίνει. Ευχαριστώ για αυτά. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάτα. Ανταλλαγή απόψεων για την επιτροπή, για τον τουρισμό. Ο, κύριος Ότουν είναι εδώ. Ο κ. Ότουν είναι εδώ, έτσι να προφέρει ο πρόεδρο. μα έδωσε αυτή τη στιγμή μια ε, πληροφορικό στοιχείο και τεκμηρίωση και ξέρετε είναι υπεύθυνο στη Γενική Διάθεση ε, και μας έδωσε αυτό το υλικό το οποίο έχουμε αναχείρας. Θα σου δώσω λοιπόν το λόγο αυτή τη στιγμή και βεβαίως να κάνετε σχόλια, ερωτήσεις όσον αφορά την παρουσίαση. Έχετε το λόγο παρακαλώ και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και είστε εδώ παρόν και μας δίνετε αφαιρετό το χρόνο σας. Ευχαριστώ Πρόεδρο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα Πρόεδρο που είμαι εδώ στη δική σας επιτροπή. Μία από τις πρώτες συναντήσεις που κάνετε και είναι καλή ευκαιρία αυτή τη στιγμή για να ξεκινήσουμε αυτή τη νέα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να σας παρουσιάσω εδώ πάρα πολύ σύντομα και να συζητήσω μαζί σας τα διάφορα αυτά θέματα. Μια στιγμή, μια στιγμή πραγματικό. Εάν θέλουν ορισμένοι να φύγουν, να φύγουν αυτή τη στιγμή και ήσυχα. Και σας παρακαλώ, εάν θέλετε να συνομιλήσετε μεταξύ σας, να βγείτε έξω να το κάνετε. Δεν θα επιτρέψω πραγματικά αυτή τη στιγμή να έχουν ad hoc ενώ υπάρχει ένας αγορητής ο οποίος έχει λάβει το λόγο. Τούτου λεχθάνους έχετε ξανά το λόγο, κύριε. Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ γιατί αυτή τη στιγμή ότι στις πρώτες αυτές συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχω την ευκαιρία να είμαι εγώ εδώ παρόν, να παρουσιάσω σε εσά και να σας κάνω αυτή την παρουσίαση την οποία και βεβαίω θα παραμείνω στα 15 λεπτά τα οποία μου παραχωρήσατε. Νομίζω πως πραγματικά είναι εκεί αυτή τη στιγμή να γνωρίζετε μερικά πράγματα. Είστε μερικοί νέοι στο Κοινοβούλιο και όχι μόνο εκεί αλλά και στην Επιτροπή αυτή υπάρχουν τρία βασικά θέματα τα οποία θα πρέπει να ξεκινήσω. Πρώτο, η οικονομική και η κοινωνική πτυχή του τουρισμού. Δεύτερο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη το θέμα που άπτεται τη ειδική τη Λισαβόνα, οι μελλοντικέ ε, ευκαιρίες καθώς επίσης και αρμοδιότητες που θα έχει η ΕΕ όσον αφορά τον τουρισμό και τρίτον παρόν και μέλλον των δραστηριοτήτων που άπτονται του τουρισμού και το οποίο εμείς το εργαζόμαστε στα πλαίσια της Κομισιόν πώς το κάνουμε και πώς αναπτύξουμε αυτές τις δραστηριότητες και ποιες είναι αυτές τις δραστηριότητες διακόπτεται όχι σταματήσω ο Βλέπω τη γραμματεία αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει αυτό το πακέτο το οποίο σας έχουν δίσει και περιμένω αυτή τη στιγμή, περιμένω τη δική σας αντίδραση όσον αφορά το πακέτο αυτήν την τεχνηρία που σας έδωσα και δείτε προς το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή για να δείξουμε πραγματικά τι γνωρίζετε για αυτά τα πράγματα και είναι μια προσπάθεια που ξεκινησε πέντε... 4-5 χρόνια πριν. Όσον αφορά την πληροφόρηση που υπάρχει εκεί, έχει την διάθεση, ε, τη διάθεση αυτή τη στιγμή και βεβαίω μπορείτε να τη θέσετε και σήμερα ή αργότερα και η δική μα μονάδα είναι ανα πάσα στιγμή στη διάθεση για περαιτέρω πληροφορίε και ερωτήσει οι οποίε θα έχετε. Πρώτον, για να ξεκινήσουμε όπω ανέφερα προηγουμένω, με το θέμα και να σας υπενθυμίσω η σημασία που έχει αυτή τη στιγμή ο τουρισμός. Δεν είναι πάρα πολύ γνωστή η διαστηριότητα όσον αφορά στις ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οπότε είναι πολύ βασική βιομηχανία θα λέγαμε το σημείο όσον αφορά την φιλοξενία η οποία γίνεται. Ξέρετε υπάρχουν τα charters, υπάρχουν ε, και εκπροσωπεί το 5% του ΑΕΠ της Ευρώπης και βεβαίως είναι το 6% της ευρωπαϊκής απασχόλησης ο τουρισμός. Αν λάβετε υπόψη επίσης και τις έμεσες βιομηχανίες, οι εργασίες οι οποίες ασχολούνται με τον τουρισμό όσον αφορά την ανοικοδόμηση, μεταφορό, μεταφορές, μέρη βέβαια όλων αυτών ε, οι θαλάσσιες μεταφορές, η ενοικοδόμηση ε, σκαφών κλπ. Φτάνουμε μέχρι το 11%. Αυτό για να σας το συγκρίνω είναι ο δεύτερος, η δεύτερη βιομηχανία, η τομέα αν θέλετε, στην ευρωπαϊκή οικονομία μετά τη διανομές. Και είναι και είναι, δύο φορές πιο μεγάλη από την αυτοκίνητο, βιομηχανία Και ακόμη δεν υπάρχει ωστόσο η αναγνώριση σε πολιτικό επίπεδο και θα μείνω σε αυτό το θέμα. Σαν τουριστικός προορισμός η Ευρώπη αλλά και διευρωπαϊκά δίκτυα και τουριστικά ταξίδια τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή από χώρα σε χώρα της ΕΕ είναι το πιο σημαντικός χώρος τουριστικής έλξης η Ευρώπη και υπάρχει κάτι ακόμη το πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είναι ότι παίρνουμε τα μη όλα τα μη, Ευρωπα... του μη ευρωπαϊκούς προορισμούς θα δηλαδή δείτε ακόμη οι Ευρωπαίοι συγκρίνεται με όλο τον κόσμο και είναι ακόμη πιο σημαντική η Ευρώπη σαν προορισμός αλλά ο τουρισμός δεν είναι μόνο σοσιοοικονομική, κοινωνικο-οικονομική επίπεδο, αλλά είναι και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής της κοινωνίας θα λέγαμε. Και θα πρέπει αυτό να έχει τη θέση που του πρέπει, αλλά θα πρέπει και τη σωστότερη διαχείριση. Διότι πρόκειται για άλλους στόχους, οι οποίες έχουν τεθεί σε άλλους τομείς, για την ανάπτυξη, την οικονομική ε, ανάπτυξη επίσης και την πρόοδο ακόμη και το 2008 όταν ξεκίνησαν αυτές οι, επι... μελέτες που γίνονται για αυτό το θέμα δείχνουν πραγματικά πως δημιουργούν απασχόληστη, βέβαια όχι της ποιότητα, αν θέλετε, είναι αυτή, αλλά συμβάλλει επίση στη συνοχή, την περιφερειακή, επίση βοηθάει πάρα πολύ στην ενίσχυση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και θα πρέπει να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι στόχοι της ΕΕ και της συνθήκης όσον αφορά το θέμα αυτό. Επ' θα πρέπει να, υπη, ε, θα ε, πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο η οι διακοπές οι οποίες γίνονται μόνο για ξεκούραση αλλά υπάρχουν και άλλες διακοπές οι οποίες είναι αν θέλετε ταξίδια τουρισμού τα οποία γίνονται και δεν είναι μόνο αυτές που είναι για ξεκούραση αυτό είναι ο λόγος για το νομίσμα και για ένα ανακεφαλαιώσω τις διάφορες πτυχές του τουρισμού στην Ευρώπη είναι ότι ποιες είναι οι αρμοδιότητες ΕΕ όσον αναφορά στον τουρισμό. Ευελπιστούμε όλοι και είμαι έτοιμο να το κάνω αυτό σε ιδιαίτερα υπό το φως των αλλαγών τα οποία θα πρέπει να γίνουν και την υιοθέτηση της, της συνθήκης στη Λισαβόνα αλλά και ήδη στην Ίκαια είναι στο ίδιο επίπεδο με την ενέργεια. Θα σοκάρει αυτή τη στιγμή, αλλά ακόμη και στην είναι στο ίδιο στο, στο 31 U ου αν θέλετε, αναφέρεται αυτό το θέμα και βεβαίω με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε αλλαγές οι οποίες γίνονται και γίνεται στην τρίτη κατηγορία όσον αφορά την ε, άθληση και θα πρέπει με, να πρέπει να γίνει πλήρω σεβαστό εφόσον υπάρχει συνθήκη του Λισαβόνος πλήρω εκ μέρου των κρατών μελών και βεβαίως υπάρχουν όροι οι οποίοι είναι πάρα πολύ ειδικοί, οι οποίοι άπτονται της ε, κοινωνικών, ε, τη κουλτούρα, του πολιτισμού κλπ. Και θα πρέπει να είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να αναλάβουμε τρο, πρωτοβουλίε με ενισχυμένη πλειοψηφία όσον αφορά αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει εργαζόμαθα στην Κομισιόν σαν να ήμασταν de facto στη συνθήκη της Λισαβόνας και υπό το φως αυτής της συνθήκης εργαζόμεθα έχετε λάβει σήμερα το πρωί ένα ολόκληρο πακέτο αυτή την εκμηρίωση που μας δείχνει ποιε είναι αυτή τη στιγμή η δική μας πολιτική τις ανακοινώσεις του Μαρτίου του 6 και του Νευρίου του 8 είναι περίπλοκα θέματα, είναι απλά και περίπλοκα βεβαίως, τα οποία θέλει να προωθήσει όσον αφορά την αηφόρο αντιγωνιστικότητα την οποία θα έχει όσον αφορά ο τουρισμός. Και φαίνεται ότι είναι ή εύκολο να γίνει, αλλά δεν είναι τόσο προφανές ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Επίσης εργαζόμαστε σε τρεις άξονες, αν θέλετε. Ο πρώτος είναι να εσωματώσουμε τον τουρισμό σε όλες τις πολιτικές ε και οποιαδήποτε ε, ε, οικονομικό εργαλείο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα έχουν πάρα πολύ σημαντική επίπτωση επί του τουρισμού και θα πρέπει να το έχουν. Πρώτη λοιπόν προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι να εξασφαλίσουμε μια πρόβλεψη όσον αφορά τον έλεγχο που θα πρέπει να γίνεται από οποιαδήποτε οργανισμό, από κράτο μέρο, από άλλη γενική διεύθυνση και έχει άπτυτε του τουρισμού. Κοιτάμε επίσης εκ του σύνεγγυς Επίσης έχουμε τον προπολογισμό έχουμε δει και έχουμε πει ότι είναι και το βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε όλα τα δημοσιονομικά εργαλεία αυτή τη στιγμή είναι προτεραιότητα για τα αγροτικά, στο ΡΑΙΦ, στο, ε, για το πρόγραμμα του Λεωνάρντου Νταβίντσι, του πλαισίου ανάπτυξης κλπ. Υπάρχει πάντα διασύνδεση και μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα οι οποίοι συνεργάζονται αγαστά για αυτό το θέμα. Δεύτερος άξονας, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι η προώθηση όσον αφορά την αηφόρο ανάπτυξη, το αηφόρο, αν θέλετε, του τουρισμού. Ξέρετε, είναι το ίδιο πράγμα και δεν είναι ένα νόμισμα με δύο, ε, με δύο όψεις. Επίσης αναπτύξουμε μία άλλες δραστηριότητε σε τρεις τομείς, δηλαδή προωθούμε μόνιμους προορισμούς, δηλαδή το βασικό προ... προϊόν το οποίο είναι ο τουρισμός είναι όσον αφορά το προορισμό. Αϊφόρος προορισμός και ο οποίος μπορεί να αναπτυχθεί στο επόμενο δίκτυο. Υπάρχουν περιοχές 16 οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι πολύ προθυμένες. Επίσης, ποιος... Είναι άλλες περιοχές οι οποίες είναι επίσης μια τρίτη η οποία με το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας όπου υπάρχουν θεματικές θεματικές, θεματικοί προορισμοί, πράγμα το οποίο προσπαθεί να δούμε ποια είναι η διαχείριση εκείνων των προορισμών που μπορούν να διαχειριστούν με τέτοια τρόπο σε τοπικό επίπεδο που να είναι αηφόρος. Επίσης, όλα αυτό το κάνουμε όχι μόνο για το περιβαλλοντική πτυχή αυτού του θέματος, αλλά στους τρεις άκρους που προανέφερα για να υπάρξει ισορροπία, μία ισορροπία μεταξύ οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντολογικού παράγοντος. Ένα άλλο όσον αφορά τον τομέα αυτόν, το περιβαλλοντολογικό, είναι να έχουμε ότι να είναι οι εταιρείε να είναι υπεύθυνε αυτό το πρόγραμμα να πτήσουμε για να μπορούν να εκπονήσουν και γιατί θέλουν πάρα πολύ την ανάπτυξη. Ξέχασα να σας πω ακόμη ότι στο δίκτυο αυτό το οποίο σας έχω πει θέτουμε μια μικρή προπαρασκευαστική εργασία η οποία γίνεται που θα ξεκινήσει, που ξεκινήσει το 9 και για αυτό το θέμα έχω δει τροπολογίες οι οποίες έχουν κάνει και βεβαίως θα περάσει αυτό αύριο στην Ψηφορία. Ε, ψηφοφορία που θα γίνει αύριο. Και το λικό είναι η, η πρόθεση η οποία θα γίνει μεταξύ των τουριστών πρέπει να είναι αυτή υπεύθυνη περιβαλλοντολογικά. Στα τελευταία δεκαετία του 90 είχε, ε, στην δεκαετία του 90 είχαμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα και έχουμε σχέση με όλη αυτή την εκμετάλλευση που μπορεί να γίνει όσον αφορά τα παιδιά, την πορνεία και άλλα τα θέματα, κατά πόσο ο τουρισμός μπορεί να λοιπόν θα μπορούσε να είναι λοιπόν υπεύθυνο. Αναπτύξαμε λοιπόν μετά την υιοθέτηση του Κοινοβουλίου μια τρίτη προσπάθεια όσον αφορά τον κοινωνικό τουρισμό στην Ευρώπη αναπτύσσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο αποκαλείται Καλυψό και εφαρμόζουμε σε αυτό το πρόγραμμα μια σειρά δραστηριοτήτων όπου υπάρχει μια καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων και σκοπός είναι να υπάρξουν ανταλλαγές μεταξύ τουριστών που έχουν ειδικά ενδιαφέροντα μεταξύ κρατών, ε, μεταξύ κρατών στην χαμηλή τουριστική περίοδο, όχι στην υψηλή. Πράγμα το οποίο όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά είναι πολλές φορές αρνητικό αυτό το κλίμα και προσπαθούμε να υπάρξει μια ανταλλαγή μεταξύ του τρίτης ηλικίας, των πολύ νέων των μεγάλων μεταξύ ε, των 65 και άνω είτε είναι ε, συνταξιούχοι είτε όχι για τους ανάπηρους και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ταξιδεύουν υπάρχουν 40 εκατομμύρια ανάπηροι στην Ευρώπη καθώς επίσης και οικογένειες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα είναι όλοι αυτοί εκπροσωπούν 50 εκατομμύρια Ευρωπαίων 150 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι μπορούν να κάνουν αυτές τις αλλαγές. Άλλη μια δραστηριότητα την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή θέλουμε να αναπτύξουμε τη γνώση και τη διαφάνεια της τουρισμού. Έχουμε οκτώ σημεία από αυτού του σημείου. Έχουμε στατιστικές οι οποίες δεν είναι ενημερωμένες. Μπορείτε να το δείτε αυτό στα αναχείρα σκήμενα τα οποία έχετε. Τα στοιχεία μας είναι του 2006 και 2007. Έχουμε πάρα πολύ καλά ενημερωθεί, λοιπόν, θα έλεγα. Υπάρχουν, υπάρχει πλήρης έλλειψη της οικονομικής ανάλυσης και δεν έχουμε καμία οικονομική ανάλυση η οποία έχει η πρόβλεψη όσον αφορά τον τουρισμό στο μέλλον. Και ιδιαίτερα είναι πολύ αδύναμη σε περιόδους αυτή σαν τη δική μας που ότι πραγματικά υπάρχει μία πτώση του τουρισμού και Ξέρετε ότι στα επόμενα 20 χρόνια θα υπάρξει ε, μείωση και των τουριστών αλλά και των εισοδημάτων και των ε, στα επόμενα 20 χρόνια που θα γίνει. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο ε, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε αυτό το, το κλίμα της πτώσης, αν θέλετε. Ξέρετε, στον Πορτό έγινε το φόρουμ υπό τη Γαλλική Προεδρία και υπάρχει μια σειρά ολόκληρων δραστηριοτήτων που αναπτύσσεται για αυτό το θέμα, για την καταπολέμηση αυτή την, της Έχουμε αυτή τη στιγμή χρηματοδοτήσει μία, ε, έναν έλεγχο το οποίο έχουν γίνει και προσπαθεί το οποίο δείχνει 25 εκατομμύρια πολιτών τι σκέπτονται και φέτος αυτή τη στιγμή υπάρχει μια νέα επιθεώρηση, ένας νέος έλεγχος ο οποίος γίνεται για να δούμε πραγματικά τι κάνανε φέτος το καλοκαίρι και τι θα κάνουν αυτό το μέχρι το πέρας χρονιάς και πώς πραγματικά μπορεί αυτό το πράγμα να προωθήσει, να προχωρήσει. Επίσης υπάρχει μια ενδιάμεση αυτή τη στιγμή εξέταση η οποία γίνεται και ξεκινήσαμε μια μελέτη ανταγωνιστικότητας και τα αποτελέσματα τα έχουμε στο τέλος αυτού του, μι, μηνός. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν και αναλύσεις θα είναι το βασικό κλειδί το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την συνάντηση, το φόρουμ το οποίο θα γίνει για τον τουρισμό εδώ στις Βρυξέλλες το ε, Οκτώβριο και όπου θα είναι ο Επίτρος Βερχόβεν και πιστεύουμε πως η βιομηχανία αυτή νομίζω θα συμπεριλάβει όλο τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ο οποίο ασχολείται με αυτή τον τουρισμό και θα είναι το μεγάλο γεγονός της χρονιάς. Ένα άλλο ασθενέ σημείο το οποίο είναι, είναι η πρόθεση της Ευρώπης μία ολόκληρη σειρά που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή στο ε, προορισμός τουρισμού από χώρες οι οποίες αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή όπως είναι η Ινδία, η Κίνα κλπ. Νομίζω πως πραγματικά πολλές ε, μέρη αυτής της βιομηχανίας τουριστική μπορούν να παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και μπορούν να προωθήσουν πάρα πολύ για τη διαφοροποίηση αυτών τουριστικών προορισμών εντός Ευρώπης για αυτούς τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται από τις χώρες που ανέφερα. Νομίζω πως πραγματικά αυτό θα επόμενη ε, τα επόμενα χρόνια. Αυτός είναι ο σκοπός, ο λόγος για τον οποίο εδώ και τρία χρόνια έχουμε χρηματοδοτήσει αυτό το πρόγραμμα. Στην Επιτροπή ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή με, ε, Ταξιδίων και συμμετέχουν πάρα πολλοί χώρες από την Αγγλία, την Ισπανία κλπ. Αυτό, αυτή τη στιγμή αυτή η Επιτροπή έχει αναμορφωθεί και έχει αποκτήσει μεγαλύτερο κύρος και νομίζω πως πραγματικά σε επόμενα μήνες και θα έχει ακόμη περισσότερο βάρος. Επίσης αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει ένα βραβείο ετήσιο το οποίο δίνεται όσον αφορά τον τουρισμό τον τουρισμό και νομίζω πως θα υπάρξει μια αυτό το βραβείο για 22 προορισμούς οι οποίοι έχουν περάσει από αυτό το διαγωνισμό όσον αφορά τη βράβευσή τους. Θα πρέπει να το έχετε αυτό υπόψη σας. Με τούτων όλων λεχθέντων θα ήθελα να πω ότι ο τουρισμός έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Υπάρχουν πολλά που είναι στραβά μέχρι αυτή τη στιγμή αλλά ο τουρισμός δεν έχει πολιτική σημασία, την, πολιτική, την πολιτική σημασία την οποία θα έπρεπε να έχει. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο θα πω ακόμη δύο πραγματάκια, τι ακριβώς κάνουμε και πώς το κάνουμε αυτό το πράγμα. Εμείς αυτή τη στιγμή προσπάθεια έχουμε 15 άτομα και 5 βοηθούς αυτή τη στιγμή στη δική μας Γενική Διεύθυνση θα πρέπει να τη με τα κράτη-μέλη, με την κοινωνία των πολιτιστών, με τις περιοχές, με τους ε, συνδικαλιστές κλπ. Όλοι αυτοί είναι πάρα πολλοί συνεργάτες και είναι μια συνεργασία η οποία θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καρποφόρος. Εργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη λοιπόν, με τους κρατικούς καθώς επίσης και άλλους μετέχοντας σε αυτή την ή μετόχους αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να δούμε ότι εξαρτώμεθα πάρα πολύ και μέχρι τούδε από τον προπολογισμό ξοδεύουμε 4 με 5 εκατομμύρια κάθε χρόνο για τα τελευταία τρία χρόνια ιδιαίτερα για τις τρεις ε, προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει και εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα αυτό Εάν το ψηφίσετε αύριο θα ήθελα να ξέρουμε έχουμε την άποψή σας και αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή όπως αυτή τη στιγμή οι προπαρασκευαστικές εργασίες οι οποίες έχουν που τελειώνουν τον επόμενο χρόνια καθώς επίσης και η Καλυψό η οποία τελειώνει το 2011 θα πρέπει να δούμε τι θα προετοιμάσουμε από τώρα για το μετά το 2011. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο στο επίπεδο των υπηρεσιών για το μέλλον είναι ότι βεβαίως θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από τη νέα επιτροπή η οποία μόλις θα εκλεγεί και πιστεύω πως το ακρόαση του νέου επιτρόπη όσον αφορά το θέμα του τουρισμού θα του θέσετε τα ερωτήματα κυρίως για να ακούσετε τι φρονή για αυτά τα θέματα και θα πρέπει ακόμη να συγχαρώ και ορισμένα αυτή τη στιγμή τα οποία έχουμε κάνει και θα πρέπει να τα δεχθούμε αυτά γιατί βρισκόμαστε σε αδύναμη θέση ωστόσο θα ήθελαμε να σταθεροποιήσουμε την, τα κονδύλια μας στον προϋπολογισμό για τις δραστηριότητες τις οποίες αναπτύξουμε μετά το πέρας αυτών των κρατηρίων θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα την οποία έχουμε μέσα στα πλαίσια της Κομισιόν και της Γενικής Διεύθυνσης και μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ λίγα αυτά τα οποία γίνονται και με πολύ υποδύναμη. Θα ιδιαίτερα θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή ότι με τη βιομηχανία που συνεργαζόμαστε θα πρέπει να έχουμε πολύ περισσότερο συντονισμό και εκπροσώπηση, ιδιαίτερα εκείνες οι περιοχές που σας ανέφερα όσον αφορά την προώθηση και βεβαίως θα θέλαμε την ενίσχυση, την εργασιών και τις συνεργασίες με εσάς εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα αυτή την Επιτροπή, τη δική σας, και πιστώ την προσοχή σας ότι υπάρχουν και άλλες επιτροπές οι οποίες έχουν επίπτωση σε, σε άλλα θέματα ε, με τον τουρισμό συγγνώμη όπως η επιτροπή των καταναλωτών υπάρχουν οι οδηγίε οι οποίες θα έρθουν επόμενη χρονιά η Ήτρα επίσης ασχολείται του εμπορίου δηλαδή όλες αυτές οι επιτροπή περιβάλλοντος, υγείας και γιατί υπάρχουν πολλοί τομεί και πολλές επιτροπές οι οποίες άπτονται και οι οποίε κατά τη ε, δική μας άποψη θα μπορούσαν να υπάρχουν τροχοπέδι ε, αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ εν πάση περιπτώσει για αυτά τα 20-25 λεπτά τα οποία αγόρισα. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Ότουν. Δεν θέλω να ζητήσω από τους ε, συναδέλφους του ΕΛΚ να λάβει το λόγο και ο Ντεγκραντές Πασκουάλ. Ευχαριστώ. Δεν θα μιλήσω για πολύ. Θέλω από, ως εκπρόσωπος ομάδας μου να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις που πιστεύω ότι θα συμφωνήσουν και οι άλλες ομάδες. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή και να καλωσορίζω τον τουρισμό ως μια ουσιαστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πρόημο βέβαια, καλύτερα να περιμένουμε να έρθει η συνθήκη της Λισαβόνας για να γίνει ο τουρισμός κοινωτική αρμοδιότητα. Είναι σίγουρο πάντως ότι αυτό το περιμέναμε πολύ τώρα, γιατί ο τουρισμός αποτελεί βασική, βασικό τμήμα των πολιτικών πολλών χωρών το να μιλάμε για τον τουρισμό ένας Ισπανός, ένας Ιταλός, ένας Γάλλος, σίγουρα μιλάμε για την πρώτη βιομηχανία στη χώρα μας. Και όχι μόνο λόγω της, σημασίας, ε, της οικονομικής σημασίας που υπογράμμισε η Επιτροπή, της σημασίας από την οπτική γωνία της δημιουργίας θέσεων εργασίας, επίσης σημαντικό σημαντική παράμετρος, αλλά από το βάθος και τη συνέπεια που έχει η ένταξή του στην κοινοτική αρμοδιότητα. Είναι σημαντικό να υπάρξει μια ενσωμάτωση των διαφόρων αντιλήψεων των διαφορετικών κουλτουρών στον τουρισμό για να λάβουμε υπόψη το πόσο θετική είναι η ένταξη των θέσεων αυτών. Το ανέφεραν ε, ήδη εδώ. Ο πρώτος χώρος προϊσμού τουρισμού είναι η Ευρώπη. Αυτό το δείχνει ότι η παλιά Ευρώπη που την αποκαλούν μερικές φορές παλιά έτσι περιφρονητικά είναι όντως πάμπλουτη σε πολιτισμό, σε μνημεία, σε φυσική ομορφιά. Νομίζω ότι είναι καιρός να εκμεταλλευτούμε και την, τα πιο συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά θέλω να τονίσω την λογική προσέγγιση της Επιτροπής. Είναι λογικό να αποτελεί η ένταξη του κοινοτικού του τουρισμού στην κοινοτική αρμοδιότητα. Είναι αναγκαίο να κάνουμε λόγο για τη βιωσιμότητα δεν είναι κάτι συγκυριακό τουρισμός αλλά κάτι μόνιμο. Οι χώρες δε που αντιμετωπίζουν, που έχουν ισχυρό τουρισμό περιλαμβάνουν και μια διάσταση κοινωνική, ε, κοινωνική συγγνώμη, που καθιστά τον τουρισμό πραγματικά κοινωνική δραστηριότητα, ιδίως στην περίοδο των διακοπών. Επιτρέπουμε έτσι την δυνατότητα κοινωνικού τουρισμού σε κάποιες ε, περιόδους, την διευκολύνουμε το ταξίδι των νέων, τη μετακίνηση των νέων, διαφυλάσσουμε την συντήρηση των ε, ε ξενοδοχειακών υπηρεσιών και υποδομών εκτός των ε, τουριστικών εποχών που αλλιώς πρέπει να κλείσουν. Όλες αυτές οι κουλτούρες λοιπόν συμβιώνουν με τον τουρισμό, συμβιώνουν με την ανάγκη διαφύλαξης και καλλιέργειας του της πλούσιας κληρονομιάς μας. Προσθέτουμε τις διάφορες γλώσσες στο τεράστιο πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης. Σίγουρα όλα αυτά μπορεί να διατηρηθούν με βάση τις πολιτικές που κατά την άποψή μου υπογραμμίζει σωστά η Επιτροπή. Σωστά τόνισε η κυρία Τικάου μια σειρά απολογιών για τον τουρισμό που θα τις υποστηρίξουμε. Θα περιμένουμε καλύτερους καιρούς όταν Θεού και Ιρλανδίας θελόντων αρχίζει να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας θα μπορέσουμε να επιτρέψουμε στον τουρισμό να αποκτήσει μια σημαντική θέση στην ευρωπαϊκή πολιτική όπως το αρμόζει. Ευχαριστώ λοιπόν για τις πληροφορίες που μας έδωσε η Επιτροπή. Σίγουρα θα έχουμε πολλές ευκαιρίες για να μιλήσουμε για όλες αυτές τις διαστάσεις ε, του τουρισμού και από πλευράς μας να τονίσω ότι είναι σημαντικό να μπούμε πρωτοπόροι στη δουλειά στον τομέα αυτό, σε όλους τους τομείς που προανέφερα. Αυτά τα λίγα και ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Δεγκράντες Πασκουάλ. Η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για την παρουσίαση και τις πληροφορίες ε, που μας έδωσε. Είναι γεγονός ότι δεν είχαμε πολλές τέτοιες ανταλλαγές απόψεων. Πιστεύω ωστόσο ότι είναι μια χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων και ελπίζω στο μέλλον να μπορέσουμε να συζητήσουμε περισσότερο για τις υπηρεσίες ε, του τουρισμού. Όντως η συνθήκη της Λισαβόνας μετά την θέση σε ισχύ της θα μας παράσχει ένα πολύ πιο γενναιόδωρο νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορέσουμε πραγματικά να δουλέψουμε περισσότερο μαζί και να συμβάλλουμε στην ενιαία προσέγγιση του τουρισμού. Έχω μία ερώτηση. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι δραστηριότητε στον τομέα του τουρισμού μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα διαφορετικά ταμεία. Είδα ωστόσο κάποιες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ λίγοι πόροι από τα διαθροτικά ταμεία για τον τουρισμό. Πολλές χώρες χρησιμοποιούν αρκετά το Ταμείο Συνοχής ή το Ταμείο περιφερειακή ανάπτυξη. Άλλε χώρε όπω η Μεγάλη Βρετανία χρησιμοποίησαν κονδύλια από το ταμειο περιφερειακης αναπτυξης αλλε χωρε οπως η μεγαλη βρετανια χρησιμοποιησαν κονδυλια απο το προγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων τόσο ώστε να βελτιώσουν τις τουριστικές υπηρεσίε. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια περισσότερα νούμερα, κάποια ποσοστά τέλο πάντων. για τους πόρους που χρησιμοποίησαν τα κράτη για να αναπτύξουν τις δραστηριότητε και τις υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού από τα, τα διευθυντικά ταμεία. Επίσης θα ήθελα να ξέρω τι θέλει να κάνει η Επιτροπή ούτως ώστε να χρησιμοποιούνται περισσότερο τα διαφορετικά ταμεία στον τομέα του τουρισμού. Επίσης, θέλω να υπογραμμίσω την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών. Θα ήθελα να σας πω ότι κάποιες πρόσφατες στατιστικές της Κομισιόν ε, για τις καταγγελίες ε, των Ευρωπαίων καταναλωτών στο, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Προστασίας του Καταναλωτή ε, διαπιστώθηκε σαφώς ότι το νούμερο ένα πρόβλημα για τον καταναλωτή είναι οι μεταφορές. Το 31% των καταγγελιών έχουν να κάνουν με τις μεταφορικές υπηρεσίες. Όπως έλεγε ο Επίτροπος κ. Σταγιάννη, είναι θετικό να βλέπουμε ότι οι πολίτες έχουν όλο ένα και περισσότερο και μεγαλύτερη επίγνωση των δικαιωμάτων τους. Ωστόσο, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι πώς λύθηκαν οι καταγγελίες που έκαναν οι καταναλωτές αυτές. Να τους ρωτήσουμε, να ρωτήσουμε τι κάνετε για να βελτιώσετε τις υπηρεσίες προς τον πολίτη. Μια τελευταία παρατήρηση. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ανάπτυξη τουρισμού χωρίς να μιλήσουμε για σωστά ανεπτυγμένη υποδομή μεταφορών. Για να, επι... για να υπάρξει τουρισμός πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Όταν πρέπει να κλείσεις ένα πλοίο, πρέπει να κλείσεις ταυτόχρονα το αεροπορικό σου εισιτήριο, το εισιτήριο του πλοίου, του τρένου και του λεωφορείου μερικές φορές. Δυστυχώς, σπάνια υπάρχει αυτή η δυνατότητα, και η κοινή δυνατότητα του να κάνει κάποιος κράτηση για όλο το ταξίδι του. Εξού και ο μεγάλος σύνδεσμος μεταξύ τουρισμού και μεταφορών και θα ήθελα να συζητήσουμε και το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σελβία. Η κυρία Σας ευχαριστώ για τις ε, την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να θέσω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Με την ερχόμενη θέση στην εφαρμογή τη συνθήκη της Λισαβόνα, αν τεθεί σε εφαρμογή το άρθρο 195, ποια μέτρα συγκεκριμένα θα προτιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι θα κάνετε δηλαδή συγκεκριμένα από πλευρά σα ποιοι θα είναι οι στόχοι σας σε ό,τι αφορά αυτά τα εκ νέου διατυπωμένα δικαιώματα. Δεύτερο στοιχείο. Μου λείπει κάπως το θέμα της αλλαγής του κλίματος σε ό,τι αφορά τον ε, τουρισμό. γιατί φυσικά θα αλλάξουν και οι αναλογίες. Αυτό έχει αναφερθεί και σε διάφορες έρευνες. Νομίζω ότι θα πρέπει να εμπαθύνουμε στον τομέα αυτό. Για να ληφθούν και τα απαραίτητα προπαρασκευαστικά μέτρα στις ε, περιφέρειες εκείνες. Όπου για παράδειγμα θα αυξηθεί η θερμοκρασία. Ο τουρισμός είναι πολύ ευέλικτος, αλλά από κάποιες άλλες απόψεις είναι και πολύ αργός και δύσκολα προσαρμόζεται. Και να περάσω τώρα σε αυτό το θέμα των παράπλευρων εποχών. Ναι, καλό θα ήταν να εφαρμοστεί ο κοινωνικός τουρισμός στις εποχές αυτές. Αλλά Δυστυχώς σε αυτές τις εποχές ο κόσμος δουλεύει. Τα παιδιά πηγαίνουν στα σχολεία. Και αυτή η μετατόπιση αναφέρεται πολλές φορές με μεγάλες ελπίδες για τον τουρισμό, αλλά στην πράξη αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες. Γιατί πολύ απλά πολλοί κόσμος δεν έχει περιθώριο επιλογής για το πότε και πού θα πάει διακοπές και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις οικογένειες με παιδιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καταδικασμένες αυτές οι προσπάθειες. Άρα νομίζω ότι στο σημείο αυτό είναι υπερβολικά υψηλές οι ελπίδες που έχουμε, γιατί πολύ απλά αυτό είναι πολύ δύσκολα εφαρμόσιμο από το μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Δεν μιλάω για τους συνταξιούχους, Μιλάω για όλους όσοι για παράδειγμα έχουν παιδιά. Τελευταίο στοιχείο, το οποίο διαπιστώνω ότι λείπει. Υπάρχουν πολύ αρνητικές εργασιακές σχέσεις στον τουρισμό. Κακοπληρωτές, κακές συνθήκες εργασίας. Και εδώ θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Γιατί για να έχουμε ποιοτικό τουρισμό πρέπει να έχουμε και εργαζόμενους που να είναι ικανοποιημένοι. Με έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το θέμα αυτό και ως φοιτήτρια εργαζόμουν στον τομέα του τουρισμού και θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολλά θέματα. Ευχαριστώ. κυρία κυρία να παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω και εγώ, να ευχαριστήσω και εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση αυτή και κατέστησε αφές ότι ο τουρισμός αποτελεί πραγματικά ένα τεράστιο οικονομικό τομέα, τον οποίο θα πρέπει να συνδυάσουμε με τις μεταφορές όντως. Συγκεκριμένες ερωτήσεις. Στην Ευρώπη έχουμε τη δημογραφική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο αλλάζει η σύνθεση του πληθυσμού, στην Ευρώπη μειώνεται ο πληθυσμός. Αυτό τι σημαίνει ότι σε κάποιους τομείς ε, ο τουρισμός θα καταστεί σημαντικός κλάδος απασχόλησης. Για παράδειγμα, στην Ήπεθρο που για παράδειγμα δεν θα υπάρχουν πολλές δυνατότητες στο μέλλον. Και είναι και μεγάλη η πολιτιστική ποικιλομορφία στην Ευρώπη. Ερωτώ λοιπόν, Μιλήσατε για τους βιώσιμους προορισμούς που θέλετε να αναπτύξετε, για δίκτυα που θέλετε να δημιουργήσετε, που θα συμπεριλαμβάνονται διάφορες περιφερειές. Ποια κριτήρια όμως θα χρησιμοποιήσετε. Μιλάτε για την Ήπεθρο ή για τομείς οι οποίοι θα πρέπει να αξιοποιηθούν πιο πολυτουριστικά από ό,τι στο παρελθόν. Δεύτερη ερώτηση σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό τουρισμό και τα άτομα με αναπηρία, γιατί και τα άτομα με την αναπηρία θα αυξηθούν ποσοστιαία σε ό,τι αφορά τον όλο ένα και μειωνόμενο πληθυσμό. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε και από πλευρά τουρισμού σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Κατά πόσο έχει αντιμετωπιστεί αυτό ως θέμα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κυρία Μάισνερ, κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχήν γιατί η Κομισιόν είναι εδώ παρούσα στη δεύτερη συνάντηση της δικής μας Επιτροπής διότι πραγματικά βλέπουμε ότι γίνεται ο τουρισμός ε, μία, ένα φλέγον θέμα όσον αφορά το, τη δική μας Επιτροπή. Και βεβαίως ετέθη πάντοτε υπογραμμίστηκε πάντοτε το θέμα αυτό του τουρισμού και πολύ καλά γίνεται και θα πρέπει να γίνει. Ήθελα ακόμη να παρέμβω εγώ για να δείξω πραγματικά τι σημασία μεγάλη έχει ο τουρισμός αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, καθώς επίσης και ποια σελήψη έχουμε. Θα ήθελα να, τους να τον ευχαριστήσω επίσης και ότι μας είπε ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε και ότι η Κομισιόν τίνει προς αυτή την τάση. Σε, ε, σχέση με τη κρίση βεβαίως θα πρέπει να πούμε πως υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολλές δυνατότητες οι οποίες μας δίνονται, αλλά για πρώτη φορά η κρίση θα πλήξει αυτό τον τομέα. Άρα διαρωτώμε κατά πόσο μπορεί αυτή, διαρωτώμε κατά πόσον η Κομισιόν αυτή τη στιγμή έχει σαν σκοπό να βγάλει τον τομέα αυτό με τα δύο αυτά στοιχεία που τα οποία ανέφερε να τον βγάλει από την κρίση. Πρόκειται για την αύξηση του εσωτερικού τουρισμού αφενός με, με τον κοινωνικό τουρισμό ή με τους στόχους οι οποίοι είναι οι κατεξοχήν ε, στόχοι, οι, οποίοι, οι προορισμοί οι οποίοι τίθενται. Και δεύτερο στοιχείο το οποίο κατά τη δική μου ταπεινή άποψη θα πρέπει να αποτελέσει μέρος των προσπαθειών μας, δηλαδή θέλω να πω ότι ο ο προορισμός Ευρώπη θα είναι η καλύτερη, η πιο ελκυστική και πιο πολύμορφη σε σχέση με τους άλλους πόλους οι οποίοι θα αναπτύσσονται για τον τουρισμό. Και ο τουρισμός θα πρέπει έχει και έχει ε, ενέχει μάλλον αυτή την κινητικότητα την οποία υπάρχει μέσα και βεβαίως αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες όπως τη Βραζιλία και λοιπά οι οποίες είναι πόλοι επίσης αλλά θα πρέπει να έχουμε και άλλη πληροφορία εκ μέρους της Κομισιόν για να γνωρίζουμε πραγματικά τι θέλει, τι απαιτεί από μας σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συνεργαστούμε ε, με τον καλύτερο τρόπο στο μέλλον. Επίσης υπάρχει η πτυχή της επαγγελματικοποίησης των διαφόρων τομέων, των διαφόρων επαγγελμάτων σε αυτό τον τομέα των ε, διαφόρων υπηρεσιών είναι διαφορετικές, είναι ποικίλε, είναι διακεκριμένες μεταξύ τους και υπάρχει βεβαίως, δεν υπάρχει ισότητα όσον αφορά τις αμοιβέ, ε, ο, ο προσωρινός χαρακτήρας, η ποιότητα η προσφερόμενη, η προσφερόμενη συγγνώμη, ποιότητα, ο εποχιακός χαρακτήρας της εργασίας αυτής. Έτσι λοιπόν η Ευρώπη θα είναι να έχει συνείδηση αυτή τη προσπάθεια όσον αφορά την κατάρτιση καθώ επίση και την απασχόληση στον τομέα αυτό το, αυτό το τομέα. Η επόμενη αγορή, κυρία Φλασό, παρακαλώ, έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ο τομέας του τουρισμού έχει τη θέση του σε μια ευρωπαϊκή πολιτική η οποία έχει σχέση και μετά την υιοθέτηση της συνθήκης της απόνωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται διότι κατά τα λεγόμενα των συναδέλφων μου είναι στο ε, είναι στο και συμμετέχει σε όλη την οικονομία της, των χωρών μας και της ΕΕ. Πραγματικά είναι ένα φυτόριο απασχόλησης υψηλής υψηλών προσόντων, μισέων και χαμηλών προσόντων ή ανύπαρξίας προσόντων. Είναι επίσης ένας τομέας ο οποίος είναι ποικιλόμορφος, πολύμορφος, δηλαδή εστιατόρια, κατασκευές, ε, ε, ξενοδοχεία, υπηρεσίες και ξέρετε οι υπηρεσίες είναι πολλές φορές μικρομεσές επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν τον οικονομικό ιστό των χωρών μας και της ΕΕ γενικότερα. Είναι σε αυτό το μέα που θα πρέπει να προσθέσουμε και το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Εγώ θα ήθελα επ' να έχουμε μια ενίσχυση όσον αφορά το συντονισμό το οποίο γίνεται μεταξύ των τοπικών αρχών και της ΕΕ γιατί πρέπει να αλλάξουν οι νοοτροπίες. Δεν συμφωνώ με τον συνάδελφο το οποίο είπε προηγουμένως ότι υπάρχουν εποχές. Υπάρχει μια συγκεκριμένη εποχή για το στον τουρισμό. Διότι υπάρχουν πολλοί τομεί στον τουρισμό. Εγώ είμαι εκλεγμένη σε μια περιοχή, εποχή, περιοχή η οποία έχει τουρισμό και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δραστηριότητε οι οποίε επιτρέπουν να έχουμε τουρισμό σε όλη τη χρονιά. Έχουμε τις διακοπές, τουρισμό, τουρισμό διακοπών, ε, εμπορικό, α, αθλητικό, ε, ε, επιστημονικό, ε, ε, ο οποίος πραγματικά αυτός ο τουρισμός μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή του χρόνου. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο φρονώ πως πραγματικά ο τομέας αυτός μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στη δική μας οικονομία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόκ παρακαλώ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Επιτροπή για την παρουσίασή της. Νομίζω ότι θυμόμαστε όλοι καλά τον προεκλογικό αγώνα και ποια ήταν οι προκαταλήψεις του πολίτη έναντι στην Ευρώπη. Ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να πετύχει αρκετά, ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί μέσω κοινών δράσεων και στον τομέα αυτό νομίζω ότι ο τουρισμός παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή ταυτότητα, αυτό που επιθυμούμε όλοι, όχι μόνο στον οικονομικό τομέα. Είναι λοιπόν βασικό καθήκον αυτό του τουρισμού και συμφωνώ με την αρχή της επικουρικότητας και της συγκέντρωση ε, της επικέντρωσης ε, στον νεανικό τουρισμό και τον παιδικό τουρισμό και σε ό,τι αφορά τον τουρισμό των πρεσβυτέρων αν θέλετε απειλείται επίσης και ο τουρισμός ε, των ατόμων με αναπηρία. Και θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχουν πρότυπα, για παράδειγμα, για τους ε, ξενώνες νεότητας, γιατί πολλές φορές μου τέθηκε το ερώτημα αυτό. Έχει κάποια Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Να πω κι εγώ δύο λόγια, κύριε Ότουν, αν μου επιτρέπετε. Κοιτάξτε, εάν θέλετε να μιλήσετε θα ήταν ε, χρήσιμο να το λέγατε νωρίτερα. Να κάνω, να απευθύνω αν θέλετε μια έκκληση για την βιομηχανική κληρονομιά. Ένα τομέα στον οποίο είμαστε αρκετά πλούσιοι αλλά τον ξεχνάμε. Υπέρ των παραλιών, των λόφων και των βουνών. Καταλαβαίνω ότι είναι όμορφε οι παραλίες, τα βουνά, οι λίμνε. ακόμη κι εγώ. Αλλά η βιομηχανική κληρονομιά υπάρχει και είναι πλούσια και που δεν την χάνει των προτεραιοτήτων που θα αρμόζε, ήρμοζε κατά την άποψή μου. Ένα άλλο θέμα που έφεξαν έφεξαν κυρίως η κυρία Τικάου και η κυρία Γιάλα Σέντερ είναι ότι θα έπρεπε στον, στην τουριστική βιομηχανία να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα όχι μόνο χαμηλών μισθών αλλά και χαμηλού επαγγελματισμού Δεν φαίνεται ότι υπάρχουν κριτήρια που, ή επαγγελματικά προσόντα που να τηρούνται κάποιοι. Κάποια κράτη-μέλη στηρίζονται σε φοιτητέ κατά τη διάρκεια των ε, σχολικών διακοπών για να τη καλύψουν τα κενά της τουριστικής βιομηχανίας. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται να δούμε όλο αυτό το κοινωνικό τομέα της τουριστικής βιομηχανίας. Το άλλο θέμα είναι η βιωσιμότητα. Το αναφέρουν, τον έφεραν διάφοροι ε, συνάδελφοι. Εγώ δεν θα ήθελα να έχουμε το εξής σενάριο. Να μην έχουν οι αγρότες νερό για τα χωράφια τους, αλλά να είναι γύρω-γύρω γεμάτο γήπεδα γκολφ με πανάκριβο και πυκνό γκαζόν. Ωραία περιοχή είναι το Αλγκάρβε, λένε κάποιοι. Εγώ θα σας έλεγα ότι ήταν ωραίο το Αλγκάρβε μέχρι ότου κάποιοι αποφάσισαν να το κάνουν ε, τουριστικό προορισμό για, κυρίως για γήπεδα γκολφ. Πόσα Πόσα γήπεδα γκολφ χρειαζόμαστε στην Ευρώπη, θα έλεγα εγώ. Το θέμα λοιπόν της βιωσιμότητας είναι σημαντικό, ιδίω για το τοπικό περιβάλλον. Κυρία Βλαστό, ε, που δουλεύει, το είπε ότι δουλεύοντας με τις τοπικές αρχές θα πρέπει να προσπαθούμε να ακούμε τις απόψεις τους και να τους λέμε κι εμείς τι, τι πρέπει να κάνουν. Αυτά. Επίσης, δεν ξέρω και περιμένω από εσά να μου πείτε. Άλλε χώρε αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με τη Βρετανία. Δηλαδή, την Παρασκευή 24 Ιουλίου που ξεκινάνε οι διακοπές διπλασιάζονται οι τιμές. Τι συμβαίνει, τα παιδιά, οι γονείς παίρνουν τα παιδιά από το σχολείο σε διακοπές ενώ τα παιδιά θα είναι στο σχολείο τους. Μήπως μπορεί να γίνει πιο λογική, πιο λογικός ο κλάδος την τιμολογιακή του πολιτική που ενθαρρύνει τους γονείς να παραβιάζουν τον νόμο. Να παίρνουν τα παιδιά τους δηλαδή από το σχολείο χωρίς άδεια. Δεν ξέρω αν αυτό είναι βρετανικό πρόβλημα ή είναι πρόβλημα πανευρωπαϊκό. Αλλά πραγματικά ανέκαθεν με εξέπλητε το ότι η κυβέρνηση μου ανεξάρτητα από την πολιτική ε, από την ιδεολογία της δεν έχουν καταλάβει γιατί φεύγουν τα παιδιά από το σχολείο και όταν τελειώνουν οι διακοπές ανεβαίνουν οι τιμές. Ξέρω ότι τα θαύματα καθυστερούν αλλά θα δούμε. Τελευταία παρατήρηση. Οι κοινωνικές διαστάσεις των εργαζομένων στον τομέα είναι τεράστιες και εγώ θα έλεγα ότι είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε και τη βιομηχανική κληρονομιά και την ε, ε, φυσική ομορφιά. Θα σας δώσω το λόγο κύριε και επειδή σας γουστάρω γι' αυτό. Ευχαριστώ. σαν του Simpsons ε, στην τηλεόραση. Τέλο πάντων, έχω μία ερώτηση. Το... Αυτή η 10 συν 5, αυτή, αυτή η ομάδα των 15, 10 συν 5 που ασχολούνται με τον τουρισμό και που αναφέρατε, έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν ένα είδος ε, δορυφορική υποδομή Θέλουμε να το κάνουμε αυτό ε, στην Τσεχία. Δεύτερο ερώτημα. Έχετε εξετάσει το θέμα των προσόντων, δηλαδή, όπως αναφέρθηκε, αν θέλεις να δουλέψεις στον τουρισμό, πρέπει να έχεις μια άδεια. Να έχεις κάποια προσόντα σε κάποιες δε χώρες και σε κάποιους τομείς πρέπει να καλύπτει, να πληρείς και κάποια ιατρικά προσόντα. Σε άλλες χώρες μπορεί να κάνεις ό,τι θες όποιος θέλει, να κάνει ό,τι θέλει όποιος θέλει. Σε κάποιες μεγάλες πόλεις η ξεναγή πρέπει να είναι πιστοποιημένη. Μήπως θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια βάση ισότιμη στον τομέα αυτό. Επιπλέον, οι κοινωνικές, οι όροι, οι κοινωνικοί όροι δουλειά στον εργαζομένων στον τουρισμό είναι κάτι που θα έπρεπε να διερευνηθεί. Το είπατε για την Αγγλία αλλά και στη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, από όσο ξέρω, βλέπουμε συχνά να δουλεύουν στον τομέα του τουρισμού άνθρωποι με πολύ, ε, σε πολύ ευάλωτες και άτυπες μορφές ε, απασχόλησης και μερικές φορές ξεκάθαρα και παράνομα μη τηρώντα την εργατική νομοθεσία. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν παράνομα, αυτό είναι άλλο, αλλά και αυτοί που δουλεύουν νόμιμα δουλεύουν με συνθήκες που δεν τηρούν την εργατική νομοθεσία. Περιβαλλοντικά στάνταρ, ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξω. Σε κάποιες χώρες υπάρχει μία τάση να βάζουμε ε, σήμανση στα τουριστικά ε, αξιοθέατα. Ξέρω εγώ ότι μπορεί να ανεβεί κάποιος με ε, καροτσάκι. Ε, ε, θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε περισσότερο αυτό. Να πούμε ότι στην περιοχή αυτή χρησιμοποιούνται για παράδειγμα ανακυκλωμένο νερό σε αυτό το γήπεδο γκολφ. Σας δίνω το λόγο λοιπόν να απαντήσετε. Αν θα θέλετε παρακαλώ να είστε σύντομος. Αλλά σας δίνω το λόγο να απαντήσετε στις ερωτήσεις των βουλευτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι βέβαιος ε, αν θα καταφέρω τρία λεπτά πριν από τις πεντέμιση να απαντήσω σε όλες αυτές τις ε, ερωτήσεις που ήταν και πολύ ευρύς. Σα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Καταρχάς ε, θα ήθελα να σας απαντήσω σε όλους Ίσως δεν μπορέσω να απαντήσω λεπτομερώς, αλλά θα μπορέσω να σας δώσω και κάποια αριθμητικά στοιχεία σε κάποιες μέλη. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Τεγκράντες. Για την ε, πολιτισμική διάσταση του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνούμε απόλυτα με την έμφαση που δίνει και ε, το είχα, το είχα σημειώσει αλλά ξέχασα να το πω. Τη διάσταση αυτή για την ευρωπαϊκή θα γίνει που είναι πολύ σημαντική για τον τουρισμό. και για τα υπόλοιπα θέματα νομίζω ότι πάνω κάτω συμφωνεί με τις θέσεις μας. Τον ευχαριστώ για την ε, ε, υποστήριξή του. Ελπίζω η Λισαβόνα να τεθεί σε ισχύ γρήγορα, κάτι που διευκολύνει αρκετά πράγματα. Για την κυρία Τικάου. Πολλά πράγματα. Τέθηκαν πολλές ερωτήσεις. Πρώτον, η χρήση και η αξιοποίηση των διευθυντικών ταμείων για τον τουρισμό. Έχουμε κάποια αριθμητικά στοιχεία για την ε, περίοδο 2000-2006. Και λαμβάνουμε επίσης και κάποια στοιχεία για από τους συναδέλφους για το e-region. Από την Γενική Διεύθυνση Regio. Και θα πρέπει να συνδυάσουμε αυτά τα στοιχεία για να δούμε τι δαπανείται στον τουρισμό. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία. Στην περίοδο 2000 με 2006 είχαμε 5 έως 7 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία ταπανήθηκαν μέσω των τεχνικών ταμείων σε project για τον τουρισμό. Δεν είναι υπερβολικά υψηλό το ποσό, το ποσό αυτό, αλλά είναι σημαντικό και αυξάνεται μάλιστα. Μας λένε οι συνάδελφοι ότι το ποσό αυτό αυξάνεται. Επιμείναμε στις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013 να ανταποκριθούμε σε όλους τους στόχους των διευθυντικών ταμείων και μας είπαν ότι θα χρηματοδοτηθούν όλο και πιο πολλά προγράμματα τουρισμού από τα διευθυντικά ταμεία. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε τα σωστά αριθμητικά στοιχεία, γιατί αυτό θα είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά και την προσαρμογή των μελλοντικών ε, προοπτικών, σε ό,τι αφορά θέματα ποιότητα, τι μπορούμε να κάνουμε. Σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, ε, θα πρέπει να ομολογήσω, όπως ξέρετε, ότι δεν είμαι αρμόδιος. Είναι η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών αρμόδια. Σε ό,τι αφορά θέματα ποιότητας, το ξέρω ότι είναι ελλειπής η ποιότητα αυτή. Το νιώθω και εγώ ως τουρίστα σε πολλές περιπτώσεις, αλλά σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία μπορούμε να λάβουμε αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες, πρέπει να σας πω ότι δεν έχω υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες στον τομέα αυτό. Επίσης υπάρχει έντονη μεγάλη συνάφεια με τις καλές υποδομές ε, τις τουριστικές σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα δυνατότητα συνδυασμού με τα τρένα, τα πλοία, τα λεωφορεία, τα αεροπλάνα. Όλα σε αυτές οι διασυνδέσεις ασφαλώς και θα πρέπει να βελτιωθούν. Αλλά ξέρω ότι αυτό θα ενταχθεί στην μεγάλη στρατηγική για τις μεταφορές το 2020. Αν δεν κάνω λάθος, υιοθετήθηκε και σχετικό έγγραφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από κάποιου μήνες. Θα ζητήσω λεπτομέρειες, ωστόσο. Θα ζητήσω λεπτομέρειες και από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Για να σα δώσω απαντήσεις. Για την Αυστριακή, για την ε, βουλευτή από την Αυστρία. Θέσατε ένα σημαντικό ερώτημα σε ό,τι αφορά την ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Τι θα κάνουμε αν, όπως όλοι ελπίζουμε, ε, τεθεί σε εφαρμογή η συνθήκη της Λισαβόνας. Να σας πω τι δεν θα κάνουμε. Γιατί αν θέλετε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να τεθεί στο μελλοντικό μου αφεντικό, στο μελλοντικό επίτροπο, ο οποίος δεν έχει ακόμα διοριστεί. Νομίζω ότι δεν είναι η θέση μου να απαντήσω. Θα ήθελα να συζητήσω με το μελλοντικό αφεντικό μου τις θέσεις αυτές. Αλλά να σας πω ότι δεν θα κάνουμε. Δεν θα εναρμονίσουμε στην τρίτη κατηγορία αρμοδιοτήτων όλους τους τομείς ε, αρμοδιότητας, ε, βιομηχανία, εκπαίδευση, τουρισμό, αθλητισμό. Σε όλα αυτά δεν πρόκειται να υπάρξει εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας. Είναι μια αρνητική αρμοδιότητα η οποία σαφέστατα διατυπώνεται στη συνθήκη της Λισαβόνας σε ό,τι αφορά λοιπόν τις αρμοδιότητες τρίτης κατηγορίας. Μπορούμε να αναλάβουμε για παράδειγμα μη νομοθετικές πρωτοβουλίες για την καλύτερη προώθηση για παράδειγμα των ευρωπαϊκών προορισμών της ε, Ευρώπης, ε, καλύτερη διευκόλυνση των ε, τουριστών σε εποχές χαμηλής σεζόν μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε δεν περιλαμβάνει ενδεχόμενη εναρμόνιση του τουρισμού σε εθνικό επίπεδο. Αυτό πραγματικά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και είμαι βέβαιος ότι ακούσατε αυτά που είπα. Υπάρχουν κάποιοι τομείς, κάποιοι όπου μπορούμε να βελτιώσουμε τις δράσεις μας και όλα αυτά θα διαλευκολυνθούν γιατί θα χρειάζεται σε επίπεδο συμβουλίου ειδική πλειοψηφία και είμαι βέβαιος ότι θα αναπτύξουμε πολλά περισσότερα σε πολύ περισσότερους τομείς. Και φαντάζομαι ότι και ο Μελλοντικός Επίτροπος ε, θα τα παρουσιάσει όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι θα τον προσκαλέσετε άλλωστε και εσείς Πρόεδρε μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του για να παρουσιάσει τα δικά του τις δικές του πρωτοβουλίες, τις δικές του προτεραιότητες γιατί ποιος είμαι εγώ να τα προβλέψω αυτά. Για την αλλαγή του κλίματος έχετε δίκιο, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Και όλα τα μέτρα αυτά για την πρόληψη του αρνητικού αντίκτυπου και την προώθηση των θετικών, αν θέλετε, διαστάσεων της ε, αλλαγής του κλίματος, η εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση των εκπομπών, Όλα αυτά εξετάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά υπάρχει και άλλη μια διάσταση, η οποία επίσης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, η τοπική και η περιφερειακή διάσταση. Εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μικρότερο αντίκτυπο. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να προωθήσουμε τους, ε, να παρατρένουμε μάλλον τους ε, προορισμούς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να σχεδιάσουν ε, τις ατζέντε τους προκειμένου να προλάβουν ε, πραγματικά αυτή την αλλαγή του κλίματος, την αύξηση της θερμοκρασίας. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα πολλές περιοχές θα είναι πιο θερμές στο μέλλον από ό,τι σήμερα. Και βλέπουμε για παράδειγμα ότι τα καλοκαίρια είναι ήδη πιο θερμά στη Νότια Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις ε, εποχές χαμηλής σεζόν. Είπατε ότι υπάρχουν περιορισμοί για όσους εργάζονται, για όσους σπουδάζουν. Αλλά έχουμε κάποιες εποχές διακοπών. Έχουμε κάποιες ε, οικογένειες με παιδιά που δεν πάνε ακόμα στο σχολείο ή για παράδειγμα ε, παππούδες με εγγόνια και επίσης είναι μεγάλο το ποσοστό των συνταξιούχων. Νομίζω ότι είναι 50, 60, 70 εκατομμύρια οι άνθρωποι που έχουν βγει στη σύνταξη. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, αλλά είναι σημαντική πηγή εισοδήματο. Αυτοί θα μπορούν να ταξιδεύουν πιο πολύ από ό,τι ω τώρα και επίσης βελτιώνεται και η υγεία του κόσμου στην Ευρώπη. Θα μπορούν να ταξιδεύουν όλο και πιο πολύ. Ε, αυτό θα αποτελέσει κρίσιμη μάζα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε αυτού του τομεί. Και συμφωνώ με αυτά που είπατε, Πρόεδρε, προκειμένου να αποφύγουμε το φαινόμενο του να παίρνουν οι γονείς τα παιδιά από το σχολείο για να ταξιδέψουν. Επίσης δεν ανέφερα προηγουμένως, αλλά περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των ημερωτικών για το πρόγραμμα Καλυψό. Υπάρχουν κάποιες συνδιασκέψεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα γίνει και μία τον Ιούνιο του χρόνου και για το 2011 και 2012 τα τελευταία δύο χρόνια του προγράμματος Καλυψό προβλέπονται τέτοιες διασκέψεις σε ό,τι αφορά το, τις εργασιακές συνθήκες. Συμφωνώ ότι σε ορισμένες περιοχές είναι αρκετά προβληματικές, αλλά ελπίζω να μην είναι πραγματικά ανυπόστατες όπως αναφέρατε. Ξέρω ότι κάποια συνδικάτα πιέζουν προκειμένου να επεκταθούν τα δικαιώματα αυτά σε όλους τους τομείς, για παράδειγμα στους ε, οδηγούς λεωφορείων και το καθεξής, αλλά αυτά τα θέματα νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν καταρχάς στην κοινωνική κλίμακα. Και αυτό φυσικά εντάσσεται και στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης των εταιριών. Οι εταιρείε θα πρέπει να φροντίζουν τη διάσταση αυτή, γιατί άλλωστε προς το συμφέρον τους είναι. Να έχουν δηλαδή εργαζόμενους με τα σωστά κίνητρα και όχι άτομα τα οποία μετά από πέντε μήνες θα φεύγουν και να, θα ψάχνουν άλλη δουλειά αυτό αφορά και την ε, ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται. Θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση της ποιότητας, ένα καλό κατώτατο επίπεδο. Στην κυρία Μάισνερ, ναι, ξέρω, λέει ο πρόεδρος, ότι σας πιέζουμε, αλλά θα μπορούσατε να κλείσετε. Ο αγροτικός ε, τουρισμός ήταν... Το πρώτο πρόβλημα του Eden πρόκειται για το μεγαλύτερο τομέα του τουρισμού αυτού. Μιλήσαμε και για το... Πρώτα για την κυρία Αγιάλα, πώς θα βγούμε από την κρίση. Ο ευρωπαϊκός τουρισμός το 90% των 380 εκατομμυρίων τουριστών είναι ενδοευρωπαϊκός τουρισμός. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο αποδοτικότητας του ευρωπαϊκού τουρισμού. Κατόπιν, ε, οι άλλοι τουρίστες που έρχονται από τρίτες χώρες ε, εντάσσονται στο θέμα της προβολής της Ευρώπης και δεν είναι θέμα μόνο της Κομισιόν αλλά και των Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού αλλά και του κλάδου. Η Ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία πρέπει να μετέχει περισσότερε δραστηριότητε προβολή τη Ευρώπη σε τρίτε χώρε. Στην κύρια Βλαστό συμφωνούμε σε ό,τι αφορά την, ε, τα προσόντα των εργαζομένων, το ρόλο των μη, των ΜΜΕ. Ο στόχος είναι ε, Πιστεύω ότι είναι δύσκολο. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν 27 κράτη 300 περιφέρειες στην Ένωση και πάνω από 300.000 δήμοι. Η Επιτροπή, η αρχή της επικουρικότητας πρέπει να παίξει ένα ρόλο. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στους 300.000 δήμους. Ε, δεν γίνεται. Οι περιφέρειες και οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές, οι ενώσεις δήμων πρέπει να συνεργαστούν στον προϊσμό Έντεν υπάρχουν ε, οι Δήμοι, υπάρχουν ήδη 70 νικητές και θα καλέσουμε και τους, τους τέσσερις φιναλίστ. Δεν μπορούμε να καλύψουμε και τους 300.000 προορισμούς, είναι σαφές. Τα στάνταρ για, τα... για τους ξενώνες νεότητας. Δεν έχουμε τέτοια στάνταρ. Αυτό είναι θέμα του κλάδου να συνεχίσει να εργάζεται με τους καταναλωστές. Δεν θα υποχρεώσουμε όμως κάτι τέτοιο. Είναι σαφής η θέση στην Επιτροπή να μην υπάρξουν ε, πανευρωπαϊκά στάνταρ. Στο... Υπάρχει ωστόσο μια πρόθεση να γίνουν σε πιο συγκρίσιμα τα στάνταρ και να ανεβούν λίγο για να καθώς και να εκμεταλλευτούμε γενικά την καλή ποιότητα των, των ευρωπαϊκών τουριστικών υπηρεσιών για να μπορέσουμε να τις επεκτείνουμε με εφελούσια στάντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να κάνουμε την Ευρώπη έναν παγκόσμιο προορισμό δηλαδή. Τελειώνω πρόεδρε. Βιομηχανική κληρονομιά. Το πέμπτο θέμα για το έντεν του 2011 είναι η αναζωογόνηση των φυσικών χώρων, δηλαδή όλων των βιομηχανικών δομών που έχουν κλείσει, ορυχεία, εργοστάσια, παλιά λιμάνια κλπ. Παλιοί, σιδηρόδρομοι, μα υπάρχουν πάρα, πολλοί, ε, πάρα πολλές γραμμές που έχουν γίνει τουριστικά μονοπάτια στην Ευρώπη. Με συγχρηματοδότηση βέβαια. TSA. Το 2001 ζητήσαμε να υπάρξει ένα πρόγραμμα ε, συγχρηματοδοτούμενο για τους, ε, ε, για τους ε, τουριστικούς ε, δορυφορικούς που δεν είχαν όμως καμία... Ε, δεν, δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον για αυτές. Αν θέλετε να σας δώσουμε τα στατιστικά στοιχεία, αλλά τα δίνει και η Eurostat. Θα σταματήσω γιατί αλλιώ δεν θα συζητήσει τα δικά σας θέματα. Ε, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν μας δώσετε πλήρεις ε, απαντήσεις. Ευχαριστούμε. Τονίσαμε την ανάγκη να ασχοληθούμε με τον τουρισμό τόσο νωρί για να ενισχύσουμε ακριβώ την διάσταση αυτή στην Επιτροπή. Ευχαριστώ για τι πληροφορίε που μα δώσετε και τι απαντήσει στι ερωτήσει μα. Λοιπόν, θα διακόψουμε και θα ξεκινήσουν οι συντονιστέ. Αν μου δώσετε όμω την άδεια να φυγώ έξω για τρία λεπτά για να φρεσκαριστώ. Αλλιώς ε, θα γίνει εδώ πέρα θα υπάρξει πρόβλημα. Θα πάω στην τουαλέτα και επανέρχομαι.